Συνάδελφοι, δεν έχει φτάσει ακόμα η πρόεδρος, οπότε με την άδειά σας να κηρύξω εγώ την έναρξη μέχρι να αναλάβει η κυρία Γκρέσλε όταν καταφθάσει με το καλό. Με 15 λεπτά καθυστέρηση νομίζω είναι αρκετή. Πραξικόπημα λέτε έκανα, ε. Κύριος Φλάνακα. Ναι, ουαλικό. Το πρώτο θέμα που είναι ουσιαστικά το 11ο, είναι ειδική έκθεση για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας και των μεταφορών. Θα γίνει ποτέ πραγματικότητα αυτή η πολιτική επιλογή. Από το ελεγκτικό συνέδριο έχει έρθει ο κ. Μπάλτσο να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, κ. Ε, Μπάλκο. Ε, ιστορικά τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ε, τις δικές τους τεχνικές προδιαγραφές για τη σήμανση στο σιδηρόδρομο. Για να ξεπεραστεί αυτό και να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος σιδηροδρόμων, ο κλάδος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισαν να ε, εκπονούν το σύστημα ERTMS για ενιαία σήμανση έτσι ώστε να ε, αντικατασταθούν όλα τα εθνικά από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Από τον προϋπολογισμό έχουν δοθεί μέχρι τώρα 1,2 δις στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στην τρέχουσα 2,7 δις εκατομμύρια ευρώ. είναι σωστός ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η διαχείριση. Αυτό εξετάσαμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον εμβαλωματική εφαρμογή, είναι patchwork, μια κουρελού, γιατί είναι πολλοί οι διαχειριστές ε, της υποδομής, πολλές σιδηροδρομικές εταιρείες ε, και δεν έχουν επενδύσει σωστά για την υποδομή αυτή. Η δε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει κλάσμα μόνο της συνολικής δαπάνης. Οι στόχοι είναι για το 2030 για το κεντρικό δίκτυο ε, και οι αντίστοιχες επενδύσεις έτσι έχουν σχεδιαστεί. Ε, γενικά για το ERTMS, ε, για το σχεδιασμό του, βρήκαμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια στρατηγική πολιτική επιλογή ενιαίου συστήματος, δεν υπάρχει συνολική εκτίμηση για όλο το σύστημα, ούτε υποχρέωση εγκατάλειψη και παροπλισμού των εθνικών συστημάτων. Μόνο ένα κράτος μέλος, ε, ε, τα οποία ε, επισκεφτήκαμε, έχει επιλέξει ένα ενιαίο σύστημα και κατάργηση του εθνικού. Για τα υπόλοιπα, το ERTMS ακόμα είναι συμπληρωματικό προς τα εθνικά συστήματα. Τέλη του 2000 16 μόνο 8% του κεντρικού βασικού δικτύου ε, των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είχε ένα λειτουργόν ERTMS. Επίσης, το τροχαίο υλικό αντικαθίσταται ε, με βραδείς ρυθμούς και γι' αυτό συνιστούμε τα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσουν το συνολικό κόστος και να συμφωνήσουν ε, σε στόχους ρεαλιστικούς, συντονισμένους και νομικά δεσμευτικούς για εγκατάλειψη των εθνικών συστημάτων. Για τις διάφορες εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο και τις σιδηροδρόμους, βασικά αυτό το σύστημα σημαίνει κόστος χωρίς να βλέπουν το όμεσο όφελος. Ε, πολλές φορές ε, οι διάφορες εκδοχές του ERTMS δεν είναι και συμβατές μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, ε, ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα, ε, έχουμε ευεργετήματα και για τις συνδρομικές εταιρείε και τους διαχειριστές του δικτύου και ως προς την δυνατότητα μεταφορών, τη χωρητικότητα δηλαδή και την ταχύτητα. Άρα χρειάζεται και εθνική ε, χρηματοδότηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Συνδυνοδομικό Οργανισμό ΕΡΑ ε, θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια και να καταργηθούν οι ασυμβατότητες. Ο οργανισμός αυτός έχει τους απαραίτητους πόρους ε, για να ανταποκρίνονται στο έργο του, στη μεγαλύτερη ευθύνη του, να παρακολουθεί στενά και να επιβάλλει την εφαρμογή του νέου προγράμματος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν και να ευθυγραμμίσουν τα εθνικά τους προγράμματα με το πανευρωπαϊκό. Και τέλος, ό,τι αφορά τη διαχείριση των ε, διαθεσίμων κονδυλίων εκτιμούμε την επένδυση συνολικά από 80 μέχρι 190 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ μέχρι τώρα είπαμε, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο η χρηματοδότηση ήταν μόλις 1,2 δις και στην τρέχουσα 2,7 μέχρι το 2020 και παρόλα τα προβλήματα δεν έχουν απορροφηθεί όλα τα κονδύλια. Για παράδειγμα, το 50% των κονδυλίων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο μεταφορών δεν έχουν απορροφηθεί και έχουν απεμπλακεί από τη συγκεκριμένη εγγραφή. Όταν κάναμε τον έλεγχο, μόνο 50 εκατομμύρια από τα 689 ε, είχαν καταβληθεί για σχέδια του ERTMS. Και τέλος, δεν πιάνουν πάντα τόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, ε, εκεί που χρειάζεται, ας πούμε, σε διάφορα δρομολόγια διασυνοριακά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονιστεί καλύτερα με τα κράτη-μέλη για να αξιοποιούνται καλύτερα τα περιορισμένα κονδύλια που διατίθεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Μπάλκο. Και τώρα το λόγο έχει η συγγήτριά μας που είναι η κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διαθέσή μα, γιατί είναι σύντομη η παρουσίαση και γενικά δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή, θα ήθελα να συνοψίσω. Να ευχαριστήσω δε και την, ε, το Εκτικό συνέδριο για την παρουσίασή σας. Μιλάμε για το αποτύπωμα των μεταφορών, για τη χρήση των ε, σιδηροδρόμων συνδερκώς και ε, θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα όλες αυτές τις ιδέες. Θα ήθελα λοιπόν να εξετάσουμε καταρχάς τον τίτλο της ειδικής αυτής έκθεσης. Μιλάμε για την πολιτική ε, θέληση, την πολιτική επιλογή, κατά πόσον θα καταστεί ποτέ πράξη η πολιτική επιλογή. Τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία ακούμε και μας παρουσιάστηκαν, ε, μας καταδεικνύουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί το κόστος ε, είναι βαρύ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα εθνικά κράτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν αποφασίσει να εισαγάγει το ERTMS δεν έκανε μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά το κόστος και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε το δίλημα αυτή τη στιγμή και σε ό,τι αφορά το πολιτικό δίλημα που επικρατεί για τις ε, διασυνοριακές τηλεδρομικές μεταφορές και επιβατών και προϊόντων δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα και τα εθνικά συμφέροντα νομίζω και οι εθνικές σκέψεις κυριαρχούν. Όλοι θέλουμε μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου. Αυτό αποτελεί πολιτικό όραμα, αλλά δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Προφανώς και θα κοστίσει πολλά χρήματα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Για να σταματήσει, για να βληθεί η διεύρυνση του ERTMS, προφανώς θα πρέπει να είναι πολλές οι δαπάνες σε ό,τι αφορά... Α, ένα συνδρομικό χιλιόμετρο το οποίο κοστίζει από 120.000 ευρώ και πάνω. Και αυτό προφανώς θέλουμε να υποστηριχθεί από τα λεφτά του φορολογούμενου και τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την επέκταση των συνδρομών αλλά και για προνόμια για τους εργαζόμενους του κλάδου, για συντάξεις και το Τουλάχιστον αυτό ισχύει σε εμάς. Επί της αρχής θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που λέει το ελεκτικό συνέδριο. Επίσης όμως, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το ERTMS αποτελεί μία απόφαση στην οποία αντιτίθεται τελικά αυτοί που την ψήφισαν και φοβούνται ε, τον ανταγωνισμό και έτσι προβαίνουμε σε προστατευτικά μέτρα. Αυτό λοιπόν, εντάξει, αν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά σίγουρα όχι εις βάρος του φορολογούμενου και ως μέλος της Επιτροπής Μεταφορών θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει απορροφήσει και τόσο πολλά χρήματα που πραγματικά θα ήθελα να υπάρξει follow-up μετά αυτή τη, αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Η κυρία Κρέσλε, σας ευχαριστώ που, για την παρουσίαση και λυπάμαι που καθυστέρησα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Η κυρία Βέρνερ, ευχαριστώ και το αλλακτικό συνέδριο και την εισηγήτρια και την Επιτροπή. Καλωσορίζουμε τη συζήτηση αυτή και είναι καλή χρονική συγκυρία για να συζητήσουμε το ERTMS. Είμαστε γενικά σε μεγάλη συμφωνία με τις συστάσεις που έγιναν. Κάποια προστατικά το 2016 και το 2017 θεωρώ ότι έδωσαν μια νέα ορμή για την υλοποίηση η οποία το παραδεχόμαστε, παίρνει πάρα πολύ χρόνο και κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα. Έχουμε όμως το τέταρτο συνδρομικό πακέτο πλέον το οποίο ισχύει και ιδιαίτερα ο τελευταίο πυλώνα δίνει σημαντικό ρόλο προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων και ε, επιτέλους υπάρχουν και σταθερές ε, και ολοκληρωμένες διατάξεις. Δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στο σύστημα αυτό το οποίο θα υλοποιηθεί και από πέρσι έχουμε και ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση. Πολύ λεπτομερές και αυτό. Και πρόσφατος μάλιστα διευκρινίστηκε παραπέραντερο με σαφή ορόσημα ποιος πρέπει να κάνει τι και πότε και Μέχρι το 2023 έχουμε θέσει το στόχο της 40% εξοπλισμού των συνδρομικού δικτύου και είμαστε λοιπόν σαφείς ε, σε ό,τι αφορά τα τρένα αυτά τα οποία θα πρέπει να μας επιτρέπουν να πάμε οπουδήποτε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά. Προφανώς ε, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ε, και πρέπει προφανώς ο κλάδος ο ίδιος να φροντίσει να είναι σταθερό το σύστημα, να υπάρχουν σταθερές και τακτικές ενημερώσεις γιατί μόνο όλα αυτά μπορούν να μειώσουν το κόστος των ε, εγκαταστάσεων των υποδομών. Κατά δεύτερον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να, εξοπλίσουν ε, τα τρένα τους με τις ε, συσκευέ αυτές και με όλα αυτά και προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και τη για συνοριακά. Έχουμε και την διαχείριση των υποδομών, το οποίο προφανώς συνδέεται με θέματα δημόσιας εκκλησίας των κρατών μελών και θα πρέπει φυσικά και οι τροχές να είναι εξοπλισμένες με συμβατά συστήματα. Και εδώ τονίζεται η σημασία του να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα, να μην λειτουργούν παράλληλα πολλά ε, ε, συστήματα και για τις μεταφορές επιβατών και προϊόντων θα πρέπει να υπάρξει μία μετάβαση για ένα ενιαίο σύστημα. Σε ένα ενιαίο σύστημα αυτό θα ωφελήσει στο μέγιστο και εδώ φυσικά έχει να κάνει και με το θέμα το οικονομικό θα χρειαστούμε διαρκή χρηματοδότηση. Δεν είναι πολιτική επιλογή, είναι μοναδική πραγματικά επιλογή για να υπάρχει ένα πραγματικά διαλειτουργικό σύστημα. Δεν ήταν πολιτική αυτή η απόφαση το ζήτησε ο ίδιος ο συνδρομικός κλάδος και τα κράτη-μέλη να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Έχετε δίκιο, είναι αργό το σύστημα σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, ανάπτυξή του, αλλά έχουμε τρεις φορές ε, το, ε, την έκταση και την απόσταση του ERTMS εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, και έτσι ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό στην ημερήσια διατάξη. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, λοιπόν, στην ειδική έκθεση παραθμών 16 για την ανάπτυξη της Υπέτρου. Ο κύριος Στεχόσκι και η κυρία Κάρνμπαχ είναι η συγκεκριτή. Ο κύριος Τσεχόφσκι να πάρει για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω σύντομα την ε, ειδική έκθεση έκθεση ε, όσον αφορά του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την ε, αγροτική ανάπτυξη, την ε, απλούστευση καθώς επίσης και τη διασύνδεση με προηγούμενες παρουσιάσεις και εκθέσεις για τους νέους γεωργούς. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων, η αποτελεσματική δαπάνη ε, είναι πάρα πολύ ε, σημαντική και οι ε, συγγνώμη, οι οικονομικοί έλεγχοι που κάνουμε αφορούν περιφερειακά και εθνικά προγράμματα και θα σας πω ποια είναι τα ευρήματά μας είναι στα αγγλικά 4L τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ ευρεία ε, και ε, κάνουν ε, πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. Είναι πολύ μεγάλα γιατί από το 2014 μέχρι το 20 είναι μία μακρά περίοδος. Τα μεγαλύτερα εθνικά προγράμματα ε, τι να σας πω, είναι πολύ λιγότερα και εδώ έχουμε 600, ε, ε, ε, συγγνώμη, 6.000 σελίδες. Ε, επίσης, ε, είναι δύο φορές ε, ε, μεγαλύτερα από τα, από τα συνήθη προγράμματα. Η Κομισιόν απαιτεί πολλά από τα ε, κράτη-μέλη. Ενδεχομένως αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά σαφώς δεν τα κατανοούν οι γεωργοί. Είναι μακροσκελής οι διαδικασίες, γιατί ο χρόνος η έγκρισης είναι πάρα πολύ μακρύς. Το τέλος του 2015 ε, δηλαδή στο τέλος του δεύτερου έτους της νέας οικονομικής ε, περίοδου ε, εγκρίθηκαν τα πρώτα προγράμματα και άρχισαν να ελοποιούνται στην αρχή του 2016. Έχουμε φτάσει τώρα στο 2017 που κάνουμε τον έλεγχο και η πρόοδος των δαπανών ήταν μονάχα 10% και ξεκινάμε επομένως με ένα 10% μονάχα να έχει δαπανηθεί. Ε, δηλαδή ε, λιγότερο ακόμα από ε, την προηγούμενη επταετία, γιατί την αντίστοιχη περίοδο τότε είχαμε 17%. Το ζήτημα είναι ότι τώρα αρχίζουμε και ε, ε, σχεδιάζουμε την μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, τις μελλοντικές ε, προγραμματικές δηλώσεις για, το, για την γεωργική πολιτική, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και ακόμα βρισκόμαστε στο 10%. Την προηγούμενη φορά οι νέες προτάσεις ε, όσον αφορά ε, την εξέλιξη των προγραμμάτων για την Ήπεθρο ε, είχε υποβληθεί αρχές του 11 και ενώ η προγραμματική περίοδος ξεκινούσε το 12. Εδώ τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου του χρόνου ξεκινάμε την πολιτική συζήτηση για το μέλλον των πολιτικών αλλά δεν έχουμε ακόμα αξιολόγηση των προηγούμενων δαπανών. Διότι οι δαπάνες έφτασαν μονάχα το 10% και βρισκόμαστε ήδη στο 2017. Ε, επίσης, ε, τρίτο στοιχείο, ε, τα προγράμματα αυτά δεν είναι καλά ε, προσανατολισμένα όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δαπανούμε κονδύλια, Έχουμε 200.000 νέους γεωργούς που πρέπει να στηριχτούν, αλλά δεν έχουμε όμως μετρήσιμα αποτελέσματα πώς να σας το πω, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην απλή ερώτηση ποιος ήταν ο αντίκτυπος αυτής της χρηματοδότησης, αυτού του προγραμματισμού, ε, για την ας πούμε ε, ανανέωση των γενεών. Τα προγράμματα ανάπτυξης της ε, υπαίθρου δεν είναι καλά προσανατολισμένα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα τις συστάσεις μας, το λέει και ο τίτλος. Θέλουμε απλούστευση ε, και ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, προς ανατολισμό δηλαδή ε, κυρίως προς τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εκτενέστερα, δεν έχουμε προβλέψει συζήτηση, μόνο μια σύντομη παρουσίαση από την εισηγήτρια την κυρία Κάντεμπαχ. Τα είπαμε και το πρωί σε σχέση με τους νέους αγρότες, θέλω να τονίσω τα ίδια πράγματα. Αν θέλουμε να είμαστε προσανατολισμένοι στο μέλλον, χρειαζόμαστε εκτενή συζήτηση, οπωσδήποτε, και με το ελεκτικό συνέδριο ακούσαμε την παρουσίαση ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο στάδιο σχεδιασμού, χωρίς να έχουμε αξιολογήσει ή να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του παρελθόντος και τα πρώτα 10% ε, ήδη έχει απελευθερωθεί των, των κονδυλίων ε, το 2017. Χρειαζόμαστε ένα έγγραφο εργασία για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά και να κάνουμε μια συζήτηση στα πλαίσια της Επιτροπής μας, πιο εμπεριστατωμένη, πιο εκτενή. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ίσως από κοινού και με παρουσία του Επιτρόπου, γιατί καλό είναι να τα πούμε στον ίδιο. Ευχαριστώ. Ε, τέλος ε, αυτού του σημείου ήταν σύντομη η παρουσίαση. Πάμε στο σημείο 13. Έκθεση αξιολόγησης του κανονισμού. Α, συγγνώμη, ξέχασα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Äh, Ο κύριος Μίλος Ευδιευθυντής της ε, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Πέθρου, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ Κυρία εκπρόσωπε του Ελληνικού Συνεδρίου, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα ε, που μας ε, δίνεται να παρεύουμε επί τη βάση αυτής της ειδική έκθεσης, την οποία η Κομισιόν ε, καλωσορίζει. Ε, ε, επί της ουσίας μπορούν να γίνουν ε, δεκτά γενικά τα ευρήματα, ωστόσο υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα αντιμετωπιστούν στην νομική, νομοθετική πρόταση για μετά το 2020. Την 29η Νοεμβρίου θα δημοσιοποιηθεί η νέα πρόταση της Κομισιόν και οπωσδήποτε λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ε, τα συμπεράσματα ε, και την αξιολόγηση του ελεκτικού ε, συνεδρίου. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε όντως κάποια καθυστέρηση για το νομικό πλαίσιο του 2014. Έχουμε βεβαίως ως Κομισιόν καταβάλει πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής, ο οποίος είναι τώρα 24 μήνες σε σχέση με τους 39 του προηγούμενου προγράμματος. Ε, ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το ποσοστό του 10% για την ε, ε, ε, χρονιά αυτή εμείς θεωρούμε ότι έχουμε 42% των χρησιμοποιημένων δαπανών όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Επίσης θεωρούμε ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων συμβάλλουμε με μετρήσιμο τρόπο στη στρατηγική του, για μετά το 2020. Υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στα ε, έγγραφα και τις ε, παρεμβάσεις και όλα προκύπτουν ε, μέσα από στενή συνεργασία των υπηρεσιών μας και μπορώ να σας διασφαλίσω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όλους τα στοιχεία του προγράμματος. Επίσης, νέα στοιχεία έχουν εισαχθεί όπως ας πούμε οι πιο αυστηρές προϋποθέσεις, ο πιο στενός ε, έλεγχος και επιτήρηση monitoring, ο σαφέστερος καθορισμός στόχων και ε, τέλος ε, η εξάντε εκ των προτέρων ερεσιμότητα που είναι επίσης κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Επίσης όλα αυτά τα στοιχεία τα βλέπουμε σε συνέργεια και σε συνοχή μεταξύ τους έτσι ώστε να παράγουν πιο καλό αποτέλεσμα και να αποτελούν και κίνητρο για τα κράτη-μέλη. Επιπροσθέτως ε, ε, χαιρόμαστε γιατί το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει το θετικό ε, του κοινού προγράμματος επιτήρησης και των κοινών παραμέτρων και δικτών. Μέσω αυτών των στοιχείων μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα και στενότερα και αποτελεσματικότερα με τα κράτη-μέλη και βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε και εν λεπτομερία τα επιμέρους στοιχεία αυτής της έκθεσης. Να σα ευχαριστώ και νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψω στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Πρόκειται μόνο για σύντομε παρατηρήσει, για παρουσιάσεις. Γι' αυτό σίγουρα θα το ξανακοιτάξουμε το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσουμε και το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευκαιρία που μα έδωσαν να ενημερωθούμε εν συντομία για την έκθεση αυτή. Και έτσι λοιπόν περάσαμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Να, να καλωσορίσουμε τον Επιτροπό Οτινγκερό, ο οποίο θα μα παρουσιάσει την ε, έκθεση αξιολόγηση για τον Όλαφ. Πρόκειται για ένα έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ανακοίνωση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα λάβουμε και την πλήρη α, έκθεση, φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσω, να καλωσορίσω και τον Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ, τον κύριο Έλετ και... και πάλι δεν μπορέσαμε να συμμετέχουμε στον διορισμό σα δυστυχώ. Και τον Γιάννη Μούλτερ ε, την, ε, από την Επιτροπή παρακολουθήσει σας. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν που είσαστε εδώ κύριε Επιτροπέ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε ε, κύριε Πρόεδρε Μούλτερ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καθήκον φιλόδοξο να μεριμνά ε, για να ενισχυθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό θα πρέπει να γίνει και προς τα έσω, μέσα και προς τα έξω. Δηλαδή στις υπηρεσίες μας και στους υπαλλήλους μας και με όλους εκείνους που παίρνουν αποφάσεις που έχουν σχέση με τα οικονομικά, αλλά και προς τα έξω με τους εταίρους μας, με τα κράτη-μέλη. Και όλους εκείνους που συμμετέχουν σε προγράμματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό αρχίζει ενωμένη από την έρευνα μέχρι και την υποδομή. Το 2017 κάναμε κάποια σημαντικά βήματα ήδη, τον Ιούλιο φέτος. Εγκρίθηκε η οδηγία για την ποινική διοξή της απάτης που στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα τεθεί σε ισχύ. Η λόγω οδηγία. Θέλω να σας ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και όλα σας τα μέλη, γιατί με τις προσπάθειές σας συνεισφέρατε αποφασιστικά σε αυτή την έγκριση. Και μόνο το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν απάγιο δικό σας αίτημα και επιτέλους το καταφέραμε. Τον Οκτώβριο το Συμβούλιο στην ενισχυμένη συνεργασία με 20 κράτη-μέλη προχώρησε και ενέκρινε ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα, το ΕΠΟ όπως ονομάζεται στα αρχικά. 17 ήταν πρώτα τα κράτη-μέλη που συμφώνησαν, στη συνέχεια 18 και τώρα 20. Ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελπίζουμε να είναι μια καλή αφιτηρία αυτή και αρχή που εν ευθέτω χρόνο να οδηγήσει σε μια γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με συμμετοχή και των 27 κρατών μελών. Τώρα καλούμαστε εμείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η συνάδελφος Γιούροβα, οι δικές μου υπηρεσίε και εγώ προσωπικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το πράττουμε ε, έτσι ώστε το συντομότερο να αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρούμε ότι θα αρχίσει το 2020 και από την 1η Ιανουαρίου 2021 με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι σε πλήρη λειτουργία για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ε, υποχρεώσεις της που απορρέουν από την νομοθεσία. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία και ε, αποφυγή απιστίας, ε, απάτης, διαφθοράς. Όχι επειδή μειώνονται οι πόροι μόνο, αλλά γιατί έτσι αυξάνεται ε, και η εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που διαφορετικά θα χανόταν. Γι' αυτό έχουμε έναν υψηλότερο, απότερο στόχο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ίδιο επίπεδο προστασίας και εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Εδώ η Όλαφ ήταν, είναι και παραμένει πρωταγωνιστής. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Το γεγονός ότι δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σημαίνει ότι χάνει το σκοπό της και το λόγο ύπαρξης η Όλαφ. Είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Και θέλω και με την πολιτική και με το οργανόγραμμα και ε, με ό,τι χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι θα έχει τους απαραίτητους πόρους η Όλαφ για να ε, διεξάγει τις έρευνες και στα 28 κρατημέλη, προσεχώς 27. Η Όλαφ, και το γνωρίζουν οι παλαιότεροι, ιδρύθηκε πριν από 18 χρόνια. Και γενικά νομίζω είναι success story η ιστορία της Όλαφ και θέλουμε να διατηρηθεί και να επεκταθεί. Το νομικό πλαίσιο ε, θεσπίστηκε το 2018 με στόχο να ενισχυθεί η Όλαφ, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία και η ανεξαρτησία, να παραμείνει άθικτη και αναλύωτη. Πρόκειται για τον κανονισμό 883 του 2013 και μετά από εννέα μακρά έτη διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων επιτέλους εγκρίθηκε. Σήμερα στρεφόμαστε προς το μέλλον και ελέγχουμε πώς θα μπορέσουμε τα μέσα που έχουμε και τις νομικές βάσεις για την καταπολέμηση της απάτης να τα μεταξελίξουμε και να τα βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπρόθεσμα στις 2 Οκτωβρίου, όπως λέει ο κανονισμός στο άρθρο 19, έκανε την έκθεση αξιολόγησης της για την ε, υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του κανονισμού 2013. Πού είναι η συνήθιση πρακτική αξιολόγησης. Και Εγκρίθηκε λοιπόν τότε και την ίδια μέρα στις 2 Οκτωβρίου υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Λάβαμε υπόψη την Επιτροπή Εποπτείας όλα αυτού, του κ. Μίλντερ και των συναδέλφων και της γραμματείας του. Έχουν έκθεση δική του, ανεξάρτητη, την οποία σας διαβιβάσαμε και σε εσά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εποπτική Επιτροπή για την επιμελή εργασία του. Τη διάβασα την έκθεση και βοήθησε πάρα πολύ στη δική μας δουλειά. Και είναι και προς το όφελος του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συμπληρώνει αποτελεσματικά τη δική μας αξιολόγηση. Πού καταλήγουμε, σε ποιο συμπέρασμα, ότι χάρη στον κανονισμό 883 του 2013 η Όλαφ και τα τελευταία τρία χρόνια είχε καλά αποτελέσματα και μάλιστα πολύ καλά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι αλλαγές που αποφασίσατε εσείς το 2013 οδήγησαν σε σαφείς ε, βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τη δεξαγωγή των ερευνών, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με εταίρους, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των προσώπων που θίγονται από τις έρευνες τη Όλαφ. Η αξιολόγησή μας όμως έχει καταδείξει και κάποιες ελλείψεις και κάποιες βελτιώσεις που χωρούν ακόμα να γίνουν. Η αποτελεσματικότητα των ερευνών είναι το βασικό θέμα. Εκτός αυτού, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού και τώρα αμελητοί χρειάζονται προσαρμογές του τρόπου εργασίας ε, του Όλαφ, έτσι ώστε να έχουμε συνέργειες, αποτελεσματικότητα και αποφυγή επικαλύψεων. Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ένα όργανο για την αποκάλυψη και δίωξη αξιόπινων πράξεων εκτός του Όλαφ. Όλαφ παραμένει ε, αρμόδιο απολύτως για τις διοικητικές έρευνας. Ε, θα πρέπει να ενισχυθούν και οι δύο υπηρεσίες όμως, αν θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο μας, κατά πολέμηση της απάτης και ένα προπολογισμό χωρίς απάτες. Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για αποκάλυψη και δίωξη αξιόπινων πράξεων είναι ε, σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της απάτης κατά τη γνώμη μας. Έτσι βελτιώνουμε και συμπληρώνουμε τη σημερινή κατάσταση. Βέβαια η παρακολούθηση ακόμα υπολείπεται. Όταν η Όλαφ αποκαλύπτει κάποιες αξιόπινες ε, πράξεις, μέχρι σήμερα εξαρτώμαστε από τις διοκτικές αρχές των κρατών μελών. Η Όλαφ είναι και παραμένει το βασικό κεντρικό ευρωπαϊκό όργανο πριν τις διώξεις διοικητικών ατασταλιών που μπορούν να ε, καταλήξουν σε απέτηση ανάκτησης. Στη δική μας αξιολόγηση λοιπόν και γνωρίζοντας ότι για τη δημιουργία της νέας αρχής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προετοιμάζει μια πρόταση για στοχευμένη τροποποίηση του κανονισμού 883 του 2013, την οποία θα προτείνουμε και θα σας διαβιβάσουμε ε, του χρόνου την Άνοιξη. Ε, σχεδιάζουμε δύο φάσεις Ξέρουμε ότι επίκενται οι ευρωεκλογέ και ξέρουμε ότι το αργότερο, την άνοιξη του 2019, θα ολοκληρωθεί η νομοθετική σας εργασία. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση, μια δέσμη μέτρων για τον καλύτερο συντονισμό ΕΠΟ και ΟΛΑΦ και για το πώς μπορούν να γίνουν καλύτερες βελτιώσεις μετά την αξιολόγησή μας και την ε, αποτύπωση της κατάστασης, της νομικής και σε απότερο χρόνο θα έχουμε μια μεγαλύτερη πρόταση για ανανέωση του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητο από την έναρξη εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που θα έχει νόημα για την όλαυση στο μέλλον. Το κέντρο βάρους που αναφέρθηκε ήδη, ένα από τα κέντρα βάρους, στο νομοθετικό πακέτο που θα προτείνουμε την άνοιξη του 2018 είναι ότι θα πρέπει να οργανωθεί έτσι η σχέση ΕΠΟ και Όλαφ ώστε να τονίζονται οι συνέρχειες και να δημιουργείται υπεραξία χωρίς επικαλύψεις, χωρίς διπλοδουλειές, όσο γίνεται αυτές να αποφεύγονται. Η ΕΠΟ και η Όλαφ είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί με διαφορετικές εντολές και καθήκοντα που αναλαμβάνουν, με διαφορετικές δομές, με διαφορετικά μέσα με μια εντολή διακριτή για τον καθένα που θα πρέπει όμως να συνδυάζεται και με την ανανέωση και αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έχει μέσα και δυνατότητες ε, δίωξης και μάλλον ε, έρευνα σε όλα που ανταποκρίνονται στην εντολή της. Είδα και τις προτάσεις Εποπτικής Επιτροπής με χαρά και βλέπω ότι σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται αυτές. Θα δούμε που υπάρχουν κάποιες διαφορές και που μπορούμε να ε, έχουμε την επικούρηση της εποπτικής αυτής επιτροπής για ε, συμπληρωματικές βελτιώσεις και με χαρά να το κάνουμε. Ουσιαστικά θα πρέπει να φροντίσουμε για μεγαλύτερη συνοχή και συνεπή εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να έχουμε ενιαίο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό διαφορές. Οι έρευνες στα κράτη-μέλη που επιτρέπεται να κάνει η Όλαφ, με τον τρόπο που γίνονται, με τον τρόπο που επιβάλλονται τα μέτρα ή πώς πλαισιώνεται η Όλαφ ή περιορίζεται από τις διοκτικές αρχές και τι γίνεται με το ποινικό δίκαιο ε, στα κράτη-μέλη και, και τις διαδικασίες, κατά πόσο μπορεί να συμμετέχει, συμμετέχει όχι Όλαφ. Εκεί θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα ενιαίο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Όλαφ αφενός και κρατών μελών αφετέρου. Και πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος κατακαιρματισμός είναι απαράδεκτος. Απέναντι σε ένα θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει και είναι αρμόδια ε, για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστούν και οι αρμοδιότητες και να ελεγχθούν όλα ε, για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Η συλλογή του ΦΠΑ, κατά την άποψή μας, αφορά και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα βαριά εγκλήματα ΦΠΑ θα πρέπει ε, βεβαίως να είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Αλλά η Όλαφ ε, έχει μια προσέγγιση διασυνοριακή και πολύ κλαδική και θα πρέπει να υποστηρίζει τα, κράτη-μέλη και τις διοκτικές τους αρχές. Αυτό θα είναι τμήμα της πρότασης που θα κάνουμε το, το χρόνο την Άνοιξη κοιτάμε και το θέμα της καλύτερη πρόσβασης από πλευρά τη Όλαφ σε πληροφορίε, σε ό,τι αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς και πώ μπορεί να επιτευχθεί αυτό σε ό,τι αφορά ε, για την, αποκάλυψη διάφορων ειδών φορολογική απάτη. Και αν αλλάχθει, λοιπόν, αν τραποποιηθεί ανάλογα το νομικό πλαίσιο, η Όλαφ θεωρώ ότι μπορεί να δραματίσει ακόμα πιο βασικό ρόλο ως φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ως ανεξάρτητος ε, διοικητικός φορέας ε, που θα θέτει πραγματικά την προτεραιότητά του στην ε, πρόληψη και αποτροπή κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων. Κλείνοντας, θα ήθελα να θίξω και κάποιες πτυχές οι οποίες συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την Όλαφ ε. και την, τις οποίες ε, και ο κύριος Μούλτερ και ο κύκλος του θίγουν σε ό,τι αφορά τις ε, εγγυήσει για τη διαδικασία και τους ελέγχους σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Όλαφ. Δεν βρήκαμε στις ερευνές μας πιστήρια για το γεγονός ότι στο πλαίσιο το σημερινό και στα μέσα που έχει στη διάθεση της η Όλαφ υπάρχουν ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ή ότι η διαδικασία είναι ανεπαρκή σε, σε οποιαδήποτε μορφή. Η μελλοντική συνεργασία μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκή εισαγγελία. σίγουρα όμω δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο αυτό. Και θα ήθελα να πω το εξή. Η Όλαφ ε, θα παραμείνει διοικητικό όργανο που θα είναι ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε δικαίωμα καταγγελία και η όλαφα θα αντρά υπό την αρμοδιότητα αυτή ακόμα και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η προσυποστήριξη αυτής και δεν θα α, είναι τμήμα των ποινικών διώξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επί του παρόντος δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή σε ό,τι αφορά το μορφωτικό πλαίσιο για τις ε, ελέγχους και για την επιτηρήση και θα υποβληθούν σχετικέ προτάσει ε, στι αρχέ του επόμενου έτου. Θεωρώ λοιπόν ότι τα θέματα αυτά και τα θέματα διαχείριση τη Όλαφ θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ε, ενό δεύτερου, πιο περιεκτικού πακέτου το οποίο θα αποτελέσει δεύτερο βήμα και θα έχει συλλέξει στο μεταξύ και τις πρώτες εμπειρίες σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Όλαφ. και είναι σημαντική η πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 3818 προκειμένου να δούμε ποιες θα είναι του κανονισμού ε, προκειμένου να έχουμε συλλέξει ήδη κάποιες εμπειρίες τις οποίες και να εισαγάγουμε στον επόμενο κανονισμό προκειμένου ε, εξ αρχής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι Όλαφ να συνεργαστούν επί σωστών και σταθερών βάσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το θεωρήσει αυτό προτεραιότητα στο πρώτο ήμιση του 2018 προκειμένου να πετύχουμε το στόχο αυτό πριν από τις ευρωεκλογές του 2019 σε ό,τι αφορά δηλαδή τον νέο αυτοκανονισμό για τη λειτουργία τη Όλαφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Λαϊκή Πρόεδρο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση τη έκθεση αξιολόγηση και για την παρουσίαση της, του οράματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης για να μας δώσει την αξιολόγηση της δικής του Επιτροπής για την έκθεση αξιολόγησης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως υπόθηκε άλλωστε και από τον ε, Επίτροπο Χότιγκερ, η Εποπτική Επιτροπή ε, έκανε ε, συστάσεις για τον κανονισμό 883 του 2013 η Επιτροπή που έπρεπε να κάνει την αξιολόγηση ε, στις αρχές Σεπτεμβρίου ε, ήταν, ε, λειτουργούσε ήδη οκτώ μήνες και στη διάρκεια αυτών των μηνών ε, είχαμε ε, την ευκαιρία να έχουμε κάποιες πρώτες ε, εντυπώσεις για τον Όλαφ, αλλά πολύ συχνά οι πρώτες εντυπώσεις είναι και οι πιο σωστές. Η Εποπτική Επιτροπή, κατά την άποψή μας, πρέπει και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, εάν θέλουμε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του Όλαφ ε, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Και επομένως μας εξέπληξε ότι ε, το γεγονός ότι η, η ετήσια έκθεση ξεκινάει ε, με αρνητικά στοιχεία για τον Όλαφα και το γεγονός ότι η Κομισιόν αποφάσισε να άρει την ασυλία του εκτελεστικού διευθυντού και μάλιστα απόφαση που πήρε μόνη της χωρίς καμία διαβούλευση. Αυτό μας εξέπληξε δεν είχαμε ε, καθόλου λάβει γνώση όσον αφορά αυτήν την απόφαση της Κομισιόν. Επίσης σημειώσαμε, και η Κομισιόν, ε, ότι ε, η εμφάνιση της Ευρωπαϊκής εισαγγελία στο προσκήνιο χρήζει περαιτέρω διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένες. Πέραν τούτου, ε, να σας πω ότι η Ελένα Φαζένα, συνάδελφός μου, θα παρουσιάσει ε, την έκθεση με την αξιολόγηση και εγώ μπορώ να πω ότι το καθαρό μήνυμα της έκθεσής μας ε, είναι ότι δεν θα πρέπει να ε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Γενικού ε, Διευθυντού ε, το κατά πόσον θα δώσει πληροφορίες στην Εποπτική Επιτροπή. Αν η Εποπτική Επιτροπή πρέπει να παίξει τον ρόλο της, τότε θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να κάνεις αξιολόγηση αν δεν έχεις τα στοιχεία. Βλέποντας, διαβάζοντας τις εκθέσεις των τελευταίων 5-6 χρόνων, χρόνων διαπιστώνει κανείς την ίδια, ε, την ίδια διαπίστωση, δηλαδή ότι η Εποπτική Επιτροπή δεν είχε πρόσβαση ε, σε όλα τα έγγραφα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία, με την άδειά σας κυρία Πρόεδρε, θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου Ελένα Φαζέντα, η οποία σε ε, εξαιρετικά πορτογαλικά θα σας τα αναλύσει όλα. Κυρίες και κύριοι ε, βουλευτές, κύριε Επίτροπε, όπως ε, ε, υπόθηκε και προηγουμένως από τον Πρόεδρό μας, είμαστε μια εποπτική επιτροπή η οποία προετοίμασε αυτήν την γνωμοδότηση για τον κανονισμό μετά από περίπου 8 οκτάμινη εργασία. Εμείς συμμετείχαμε σε αυτήν την άσκηση την οποία θεωρούμε θεμελιώδου σημασίας και η οποία έδωσε, μας έδωσε την δυνατότητα να δούμε, να έχουμε μια ε, καλή συνολική έποψη όσον αφορά ε, την λειτουργία της ε, Επιτροπής και τη λειτουργία της Όλαφ. Υπάρχουν στοιχεία βεβαίως τα οποία ε, προφανώς ε, ε, περιλαμβάνονται εις τις αρμοδιότητες της Εποπτικής Επιτροπής που μεριμνά για την τηρήση της ανεξαρτησίας του Όλαφ. Κοιτάξτε, ε, έχουμε προβληματισμούς όσον αφορά ε, την διάρκεια των ερευνών, την προστασία των στοιχείων των ε, υποέρευνα ατόμων, αλλά και όσον αφορά το συμβουλευτικό ρόλο του Γενικού Διευθυντού. Σε αυτά τα πλαίσια η Εποπτική Επιτροπή ε, ε, εκπώνησε την γνωμοδότησή της, λαμβάνοντας ε, ως προτεραιότητες τα στοιχεία τα οποία εν συντομία θα αναφέρω. Υπάρχουν τέσσερα κεντρικά στοιχεία όσον αφορά τις έρευνες, την επιτήρηση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο μέλλον και όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στον Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις έρευνες, έχουμε υποβάλει τα εξής ερωτήματα. Το, τα νέα εργαλεία και οι νέες αρμοδιότητες ε, του ε, Όλαφ βάσει του κανονισμού 883 δίνουν την δυνατότητα στον Όλαφ να αντιμετωπίσουν ε, οποιασδήποτε παραβάσεις, απάτη ή οτιδήποτε αντιτίθεται εις ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την επιτήρηση, την εποπτεία, οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Η ε, ανεξαρτησία του Όλαφ με τον νέο κανονισμό θα διασφαλίζεται ή η νέα θητεία έχει αποδείξει αποδυναμωθεί λόγω της νέας ε, εντολής. Η Εποπτική Επιτροπή ε, μπορεί να διασφαλίσει ε, την ε, ε, ανεξαρτησία του Όλαφ, έχει την δυνατότητα να ενισχύσει τον Όλαφ εις την εκτέλεση των καθηκόντων του έτσι όπως τα έχει αναλάβει βάσει, των, βάσει της εντολής που έχει λάβει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, προστατεύονται ε, τα δικαιώματα, υπάρχουν μηχανισμοί για την ε, ε, σαφή και ορθή εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων. Επίσης, το μέλλον, πώς θα προκύψει η ανάγκη αναθεώρησης των κειμένων, πώς θα αλλάξει η δομή του Όλαφ. Η Όλαφ θα πρέπει να παίξει κατά κάποιο τρόπο ένα διπλό ρόλο ε, εάν και εφόσον ε, υπάρξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος της Όλαφ δίπλα ε, και σε συνέχεια με την, και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις έρευνες, εμείς είπαμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ομοιογενούς ερμηνείας και εναρμονισμένης ερμηνείας όλων των στοιχείων αναφερόμαστε εδώ και στους εσωτερικούς κανόνες που θα πρέπει να είναι, ε, να γνωστοποιούνται και προς τα έξω. Επίσης, ε, ο Όλαφ ε, θα πρέπει ε, να παρουσιάζει και τις ε, δραστηριότητες του εν είδη κώδικα, ενός κώδικα που αφορά ακριβώς τις δραστηριότητες του. Αλλά παρόλα αυτά να έχει τη δυνατότητα και ο Γενικός Διευθυντής να προχωρήσει σε κάποιες ειδικέ διατάξεις. Όμως δίνεται με τον τρόπο αυτό πολύ μεγάλη, υπερβολική κατά την άποψή μας, ε, υπερβολική διακριτική ευχέρεια εις τον ε, Γενικό Διευθυντή. Εμείς έχουμε στην διάθεσή μας ε, μία σειρά 28 άρθρων ε, του 2013 ε, που διαρκώς ε, όμως δεν, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουν ενταχθεί σε ένα πιο ολοκληρωμένο, ενσωματωμένο πλαίσιο. Πρόκειται δηλαδή για άρθρα ξεκάρφωτα, μεμονωμένα, τα οποία σίγουρα δεν μπορούν να εγγυηθούν την προστασία των δικαιωμάτων, αλλά ούτε καν την αποτελεσματικότητα αποτελεσματικότητα των ερευνών ε, θα πρέπει να καθοριστούν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για τις έρευνες. Όσον αφορά την εσωτερική δομή του Όλαφ, ε, ε, διαπιστώσαμε ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Η μονάδα η οποία ε, η ίδια η ομάδα είναι αυτή η οποία αποφασίζει την πρόθεση της έρευνας και αυτή που αποφασίζει για το κλείσιμο ε, της ε, έρευνας. Θα πρέπει όμως να ελέγχεται η νομιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία χρησιμοποιούμε διαφόρους εμπειρογνώμονες στα πλαίσια του Όλαφ έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα οι έρευνες Επίσης, στον ε, κανονισμό θα πρέπει ο νομοθέτης να δείξει ποιες είναι οι κύριες, τα κύρια πεδία, η γεωργία, τα τελωνία κτλ. Ε, στα οποία ε, μπορεί κανείς να ε, έτσι ώστε να γίνουν καλά οι έρευνες. Η, η δομή κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι τέτοια που θα ενισχύει την ανεξαρτησία του Όλαφ. Ε, Α θυμηθούμε λίγο βασικές αρχές ε, του ε, ανοίγματο μια έρευνα. Όντω, θα πρέπει αυτή να είναι απολύτως ανεξάρτητη και να μην δέχεται καμία πίεση ή υπόδειξη από εθνικές αρχές ή οποιασδήποτε άλλες αρχές. Ακόμα και απόφαση του Γενικού Διευθυντή για μη ύπαρξη έρευνα, θα πρέπει να κοινοποιείται με την σωστή αιτιολόγηση έτσι ώστε να να μπορεί ε, ε, να ενισχύεται η ανεξαρτησία του Όλαφ. Πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, και ε, οι οποίες προϋποθέτουν βεβαίως ε, την απλήρη ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντού. Όσον αφορά την περίοδο των ερευνών θα πρέπει βεβαίως να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και πολλά άλλωστε εργαλεία ήδη είναι διαθέσιμα πρέπει ε, να καταβληθούν προσπάθειες για τη σωστή διενέργεια των ερευνών. Ε, ε, είναι γνωστό ότι ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, ισχυρό έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η ερευνητική διαδικασία. Όσον αφορά την διάρκεια των ερευνών θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι έρευνες σε λογικό χρονικό διάστημα ανάλογο με την περιπλοκότητα ε, της ε, κάθε υπόθεσης. Αυτό είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό. Και βεβαίως οι έρευνες μπορούν να προχωρήσουν μόνο εάν και εφόσον όλα τα στοιχεία γίνονται γνωστά και δημοσιοποιούνται, πράγμα που όπως είπε και ο Διευθυντής προηγουμένως ε, δεν ισχύει. Η δυνατότη, ε, θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα τροποποίησης αυτών των ε, διατάξεων πάνω σε συνεργασία και με την Εποπτική Επιτροπή. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Όσον αφορά το κλείσιμο των ερευνών, έχουμε διαπιστώσει ότι σε ένα πλαίσιο στο οποίο 50% των υποθέσεων δεν έχει προχωρήσει, των συστάσεων μάλλον, ε, ε, και βάσει ε, της, ε, ε, των εμπειριών που έχουμε, αυτό, ευθύνεται, αυτό βασι, οφείλεται σε πολλά στοιχεία. Ενδεχομένως δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, έχουν παραγραφεί τα δικήματα ή οτιδήποτε. Λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει η αρχή του, της, του ελέγχου εξάντε Ε, εμείς ε, βάσει της έρευνάς μας ε, είδαμε ότι η Επιτροπή Επιτήρησης έχει τη δυνατότητα να να βοηθήσει ε, στην άσκηση των καθηκόντων του τον Γενικό ε, Διευθυντή ε, και βεβαίως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όταν ανοίγει μια έρευνα να κοινοποιείται δεόντως και στις δικαστικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Είναι σημαντικό να αποστέλλονται ε, όλες ε, οι πληροφορίες. Θα πρέπει να δίνονται ε, όλα τα στοιχεία στην Επιτροπή Επιτήρησης. Να δεσμεύεται επομένως ο Όλαφ απέναντι σε αυτήν την Επιτροπή και να απαντούν σε κάθε περίπτωση ε, όλες τις πληροφορίες ε, χωρίς να μπορούν να αρνηθούν ή να αγνοήσουν τα αιτήματα αυτά. Είναι ε, εξαιρετικά σημαντικό αυτό το τελευταίο στοιχείο. Βεβαίως η Επιτροπή Επιτήρησης έχει πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει. Η Πρόεδρος ζητάει από την ομιλήτρια να μην μιλάει με τέτοια ταχύτητα. Έλεγα λοιπόν ότι το γεγονός ε, ότι ο Γενικός ε, ε, Διευθυντής αποτέλεσε αντικείμενο νομικής, δικαστικής συγγνώμη, διαδικασίας και έρευνας από τις βελγικές αρχές μας προβληματίζει πάρα πολύ και θέλουμε να κατανοήσουμε και αναρωτιόμαστε πού οφείλεται αυτή η κατάσταση και πώς μπορεί να αποφευθεί στο μέλλον τέτοια μια αντίστοιχη κατάσταση. Θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να ε, δίνονται όλα τα απαραίτητα εχέγγυα. Ο κανονισμός, ε, κατά την άποψή μας, ε, θα πρέπει να αποφύγει να δώσει την δυνατότητα να παρουσιαστούν αντίστοιχες καταστάσεις και περιστάσεις στο μέλλον μέσω της σύστασης μηχανισμών ελέγχου και επιβεβαίωσης, εξακρίβωσης της νομιμότητας ε, και μάλιστα τα εργαλεία αυτά, οι μηχανισμοί αυτοί να είναι πολύ σοβαροί. Η Επιτροπή Επιτήρησης ε, θεωρεί ότι ο νομοθέτης ε, θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο για την κάλυψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και την κάλυψη της ορθότητας των διαδικασιών. Ε, όσον αφορά το μέλλον, τις ε, σχέσεις ε, του Όλαφ με την μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως έχει οριστεί από τον κανονισμό του προηγούμενου Οκτώβρη, εδώ αναμειγνύονται ενεργά και τα κράτη-μέλη και επομένως ξαναγυρνάμε στην αρχική ερώτηση. Μέχρι ποιο βαθμό θα απαιτηθεί αναθεώρηση του κανονισμού και επίσης η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ποιο τρόπο θα, και μέχρι ποιο βαθμό θα επιδράσει, ε, θα έχει επιρροή ε, στην διάρθρωση και την, ε, τις αρμοδιότητες του Όλαφ εμείς θεωρούμε ότι όλες, ε, ε, όλα τα θεσμικά όργανα ε, θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους και να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι η εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και βεβαίως εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε. Αλλά με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει όλα σε, αυτό το, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, σε αυτό το νέο ε, περιβάλλον, θα συνεχίσει ε, με τον ίδιο τρόπο να εργάζεται, θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες όλα, θα πρέπει να αξιολογεί κάθε διαδικασία πριν αυτή προωθηθεί προς την Ευρωπαϊκή ε, Εισαγγελία λόγω της απέτησης η οποία ε, υπάρχει βάσει των ε, ε, νομικών κειμένων και βάσει της εντολής. Θα πρέπει επομένως να από την άλλη πλευρά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ζητήσει τα ενδεχομένως και στο μέλλον ε, κάποιες, ε, ε, να αναλάβει το τμήμα των διαδικασιών στα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν δεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα, σε ορισμένες χώρες δηλαδή ο Όλαφ θα παίζει στην ουσία το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και θα πρέπει να δούμε ε, ε, ε, και όλα αυτά πάντα όσον αφορά τον έλεγχο των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που η Όλαφ διατηρεί τις διαβριμένες αρμοδιότητες, είναι φυσιολογικό ότι ε, οδηγούμαστε να πούμε ότι οι λειτουργίες της Επιτροπής ε, ε, είναι ακόμα σκόπιμες και δόκιμες και επομένες και επομένως θεωρούμε ότι πραγματικά θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες επί τη βάση των οποίων θα γνωμοδοτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της γνωμοδότησης αυτής. Ιδού, λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον και καθόλου χαρμόσυνο. Δύο γραμμές δηλαδή. Η Εποπτική Επιτροπή ασχολήθηκε εκτενέστατα και περιστατωμένα με τη μελέτη αξιολόγησης και θεωρεί, κύριε Επίτροπε, ότι χρειάζεται πολύ ευρύτερη αναθεώρηση του κανονισμού από ό,τι προτείνετε εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα έγγραφά της. Τώρα τι θα κάνουμε, αν κοιτάξουμε τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει 120 άρθρα. Και ο κανονισμός Όλαφ είναι φτωχό συγγενής. Ο αρχικός κανονισμός είχε μόλις 14 άρθρα. Τώρα το διπλασιάσαμε ας πούμε. Αλλά δεν είναι επαρκές αυτό για τις επιπτώσεις που έχουν στις ζωές και των ανθρώπων και τις σταδιοδρομίες των υπαλλήλων τέτοιες διοικητικές έρευνες. Όλαφ. Άρα μήπως να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αν κοιτάξουμε ε, τον κανονισμό ΕΠΟ και το συγκρίνουμε με την Όλαφ, ήμουν τότε εισηγήτρια ε, και ε, ε, γνώρισα αντίσταση και από το Συμβούλιο και από τον πρώην Γενικό Διευθυντή του Όλαφ, ε, γιατί ήθελα να παρέμβω άμεσα. Αν δεν κόψουμε τώρα αυτό τον κόμπο, θα χάσει και δυνατότητες λειτουργίας η Όλαφ και θα φύγουν και από το δικό μας έλεγχο και της δικής σας αρμοδιότητας και της Εποπτικής Επιτροπής. Είναι παγόβουνα αυτά ε, που βρίσκουμε. Δηλαδή βλέπουμε με την κορφή του παγόβουνου, δεν μας αρέσει αυτό που βρίσκουμε και μετά δεν μπορούμε να αγγίξουμε όλο το άλλο που είναι βυθισμένο. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία που δεν μπορούμε εμείς να τα ε, θεωρούμε ικανοποιητικά και υπάρχουν και νέες υπόνοιες και νέες υποψίες και αποχρώσεις ενδείξεις και περισσότερα παγόβουνα από ό,τι θα θέλαμε. Και επειδή δεν θέλω εγώ να χαθώ εκεί στον πάγο, ε, χρειάζεται θαραλέα μεταρρύθμιση για να λύσουμε τα προβλήματα και κάποια πράγματα να τα πούμε με το όνομά τους. Η εισαγγελία ευρωπαϊκή έχει checks και balances, εσωτερικούς ελέγχους και εξισορροπήσεις ε, και αντίβαρα. Αυτό η Όλαφ δεν το διαθέτει και είναι και προς το συμφέρον τους να λυθούν τα προβλήματα της ε, διακυβέρνησης το δικαίωμα ελέγχου. Τα ίδια προβλήματα έχει και έκθεση αξιολόγηση. Τα λέει το έγγραφο τη Επιτροπή, σελίδα 10, ότι κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να τα πούνε ε, με βεβαιότητα γιατί δεν είχαν ε, πρόσβαση στα στοιχεία. Και δεν μπορούσαμε να συνδέσουμε ε, ορισμένα αποτελέσματα με κάποιες έρευνες λόγω του κανονισμού. Θα πρέπει να έχουμε τώρα το θάρρος να τα πούμε έξω από τα δόντια. Και να ελέγξουμε ε, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς ε, φόβο και πάθος, ας πούμε, τον τρόπο λειτουργίας της όλα. Αυτά είπατε εσείς, κύριε Επίτροπε. Πώς μετράμε την ε, αποτελεσματικότητα στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρώσει και τις υποθέσεις με συστάσεις, δηλαδή που έχει βγει και κάτι. Τότε, ε, κατά μέσο όρο, είναι 50 με 60%. Το έτος 2012 και 2016 ε, ήταν κακές χρονιές. Το 2012 είχαμε 31% και το 2016 43%. Ήταν οι χρονιές που είχαμε κατά ποσοστό ε, τα χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις υποθέσεις που είχαν ανοίξει. Έχει πρόβλημα επιτυχίας όλο και ολοκλήρωσης των υποθέσεων. Και έχετε δίκιο και εσείς και η αξιολόγηση, γιατί δεν έχει κάποια δικαιώματα ε, όλα για να προχωρήσει. Αλλά με τη νομική βάση που έχουμε και τις δυνατότητες ελέγχου εξωτερικές και εσωτερικές και την έλλειψη εσωτερικών ελέγχων και αντιβάρων, έχω πρόβλημα. Ας πούμε, πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα. Αν δεν βελτιωθεί η διαχείριση, εγώ έχω μεγάλες αναστολές να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και για τραπεζικά δεδομένα και οι θυγόμενοι από τις διαδικασίες και τις υποθέσεις αυτές θα είναι εκτεθειμένοι σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί έχουμε προβλήματα με το νόμιμο και το νομότυπο ορισμένων διαδικασιών. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν πριν προχωρήσουμε στα επόμενα. Και σας ενθαρρύνω κύριε Επίτροπε. Πολύ ενδιαφέρουσα η γνωμοδότηση της Επιτροπής, της Εποπτικής και σας ευχαριστώ πολύ ε, είπε σε λεπτομέρειες ότι ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει πολύ σύντομα να γίνει νομοθεσία. Αυτό είναι θέμα του νομοθέτη, όχι του Γενικού Διευθυντή εντολές προς ε, υπαλλήλους. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εδώ και 18 χρόνια έχουμε τα ίδια προβλήματα. Γιατί έχει διτό χαρακτήρα η Όλαφ. Από τη μια είναι η διοικητική διερεύνηση και από την άλλη η ποινική. Δεν θα ήταν καλύτερο ο Όλαφ να γίνει αμυγός διοικητικό όργανο για διοικητικές έρευνες και θα βοηθούσε να έχουμε ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να συγκρίνει τα κράτη-μέλη. Τι δικαιώματα έχουν κάποιες κρατικές αρχές που κάνουν διοικητικές έρευνες, τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις. Έτσι ξεκίνησε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήταν πολλά υποσχόμενη αυτή η οδός. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για να αρχίσουμε να νομοθετούμε. Αν δούμε τι λέει ο κανονισμό για την εισαγγελία, έχω μεγάλα προβλήματα και μεγάλη δυσκολία να καταλάβω πώς όλα αυτά θα μπουν ε, σε ένα βλάκι. Ας πούμε, για να γίνει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ε, θα πρέπει να ξεκινήσει μόνο εφόσον η προοπτική φυλάξη είναι άνω των 4 ετών, η ποινή που προβλέπεται. Στον Όλαφ δεν λέει τίποτα τέτοιο. Γιατί γίνεται ε, όταν ε, έρχεται η εισαγγελία και ζητάει από τον Όλαφ δικαστική συνδρομή ή να είναι κάποια αξιόπινα ε, αξιόπινες πράξεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Όλαφ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πολύ συγκεκριμένες ε, επίσης εντολές για το πώ διαβιβάζει δεδομένα, ενώ όλα όχι, που μπορεί να έχουν σημασία ποινική. Ή κάποιος που διερευνάται από την Όλαφ δεν έχει επουδενή το δικαίωμα να ε, έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, στις διαδικασίες. Τουλάχιστον σχόλια να κάνει για τις διαπιστώσεις Όλαφ. Αυτό είναι στην ποινική δικαιοσύνη βασικό ε, δικονομικό δικαίωμα. Στη διακητική διερεύνηση είναι αλλιώ. Στην εισαγγελία έχει πλήρη γνώση του φακέλου και της δικογραφίας, ας πούμε, ο ε, ενδιαφερόμενος, ο οποίος ερευνάται. Είναι πολύ ευρύτερη λοιπόν η κάλυψη που έχει η εισαγγελία από ότι Όλαφ αν όλα αυτά δεν ευθυγραμμιστούν, κινδυνεύουμε να χαθούμε σε τριβές και σε απόλυση ακριβώς από τη σύγκρουση αυτών των διατάξεων. Θα πρέπει ε, να λυθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει μόνο ένα άρθρο στον κανονισμό ε, για την εισαγγελία που αναφέρεται σε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τον Όλαφ. Όλα αυτά που σας λέω όμως δεν αναφέρονται καν, για να μην πω ότι προτείνεται και τρόπος να λυθούν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι και όλα φυσικά έχει κάποια προβλήματα. Ακούμε ένα σύστημα case management, 9 εκατομμύρια ευρώ και θέλουν άλλα 5 εκατομμύρια να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο τα ζητούν αυτά. Γιατί ακούμε ότι υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας και τα συστήματα αυτά και τα περιεχόμενα μπορούν να αλλάχθουν χωρίς τεκμηρίωση. Αυτά τα πράγματα είναι δραματικά που μειώνουν και, την, και αφορούν την αποτελεσματικότητα του Όλαφ και τη δυνατότητα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι λοιπόν πολλά τα προβλήματα. Προσπάθησα να τα θίξω λίγο επιγραμματικά και να πω στην Επιτροπή μας ήδη ότι θα κάνω ένα έγγραφο εργασίας βάσει της γνωμοδότησης, βάσει του κανονισμού για την εισαγγελία να βλέπουμε τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και βάσει της αξιολόγησης, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, να κάνουμε μια απογραφή και μετά καλά θα κάναμε πραγματικά να ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει κάτι παραπάνω από το ελάχιστο. Μας είπατε προηγουμένως κύριε Επίτροπε ότι χρειάστηκαν εννέα χρόνια. Αφαιρέστε τα τέσσερα όμως γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πανημέλα πρόταση και μετά την πήρε πίσω. Δύο φορές το έκανε αυτό, μετά τρίτη πρόταση. Δηλαδή χάσαμε πάρα πολύ χρόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αμφιταλαντεύεται. Το ξέρω ότι διαφωνούσατε ε, για το τι πρέπει να γίνει. Είναι δύσκολο το πράγμα. Τώρα όμως ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να συντονιστούν τα δύο όργανα, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα δούμε την όλη ιστορία όλα αυτά να επαναλαμβάνεται που ήταν μια ιστορία η οποία δεν ήταν και τέλεια. Ούτε μπορεί να μας ικανοποιεί και δεν μας ικανοποιεί. Έχουν ζητήσει συνάδελφοι το λόγο τέσσερις. Πρώτος ο κύριος Γιάβορ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Έτενγκερ και την Επιτροπή για την αξιολόγηση του κανονισμού και συμφωνώ με πιο πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην έκθεση αυτή. Ιδιαίτερος δε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να ευδηρηθεί ο ρόλος της Όλαφ ε, ακόμα και μετά την σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ιδιαίτερος ε, επειδή κάποια κράτη-μέλη δεν θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ως εκ τούτου ο Όλαφ παραμένει το βασικό ερευνητικό σώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερο έλεγχο των δαπανών στα κράτη-μέλη, αλλά επίσης επειδή τα κράτη-μέλη τα οποία θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρώ ότι θα έχουν ε, προστιθέμενη αξία με την Όλαφ. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι εντοπίστηκαν ε, κάποια προβλήματα, κάποιες ατασταλίες σε ό,τι αφορά τις έρευνες που έγιναν. Και νομίζω ότι οι έρευνες της Όλαφ ε, να βασίζονται στην εθνική νομοθεσία είναι κάτι απαράδεκτο, το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε με διαφορετική νομική δάση, δηλαδή να κάνει τις έρευνές του ΟΛΑΦ αυτα αυτά, διάφορα κράτη-μέλη, αυτό θα πρέπει σίγουρα να το κοιτάξουμε. Και Επίσης, συμφωνώ ότι η εντολή και η ερευνητική αποστολή του όλα αυτά πρέπει να διευρυνθεί σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στην τον εντοπισμό παραχάραξης ε, και προϊόντων ε, πλαστών. Ε, ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα προβλήματα και συμφωνώ με την κυρία Κρέσλε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί βαθύτερη μεταρρύθμιση του Όλαφ, καθότι υπάρχουν κάποια θεμελιώδη προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε, αλλά να προσθέσω και κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι είναι κρεμή ακόμα ω ερωτηματικά. Ε, ανέφερε και η κυρία Φαζέντα το θέμα ε, του follow-up των συστάσεων του Όλαφ. Συμφωνώ, δεν μπορούμε να προσμετρούμε την αποτελεσματικότητα του Όλαφ μόνο με αριθμητικά στοιχεία, με τις υποθέσεις που ανοίγουν. για τη τελική ανάλυση η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Όλαφ έχει να κάνει με το κατά πόσο ακολουθούνται οι συστάσεις από τα κρατημέλη και κατά πόσο ε, πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Γίνονται, για παράδειγμα, έρευνε από τις εθνικές ε, αρχές και συχνά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και συχνά ο Όλαφ δεν έχει καν πληροφορίες. Δεν ενημερώνεται καν για το ποιες από τις συστάσεις του ακολουθούνται από τα κρατημέλη. Προφανώς λοιπόν αυτό ε, δεν μας επιτρέπει να προσμετρήσουμε την πραγματική αποτελεσματικότητα. Δεύτερο στοιχείο, η διαφάνεια των συστάσεων του Όλαφ. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το ζήτημα αυτό, και ξέρω ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι στάσεις του Όλαφ αποστέλλονται στις εθνικές αρχές και δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Και προφανώς και οι ποινικέ διώξεις ε, επιτάσσουν μια κάποια εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά τα έγγραφα. Από την άλλη φυσικά έχουμε και το συμφέρον του πολίτη και το δικαίωμα του πολίτη να έχει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Συμπεριλαμβάνομαι ένα εκτό συστάσεων. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σαφή ρύθμιση αυτού. Σε κάποιες περιπτώσεις δημοσιεύονται οι συστάσεις του Όλαφ από τα κρατημέλη, από τις κυβερνήσεις. Σε άλλε περιπτώσεις όμως δεν υπάρχει τρόπος να έχει κάνει πρόσβαση στις συστάσεις αυτές. Και αυτό θεωρώ ότι πραγματικά υπονομεύει την σταθερότητα του συστήματος και είναι πολύ διαφορετικές οι προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των συστάσεων του Όλαφ. Θα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ του απόρριτου και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ε, ποινικών ε, ε, διώξεων και ερευνών και τη δικαιώματο πρόσβαση σε... στα έγγραφα αυτά, στι συστάσει αυτέ. Τρίτο ζήτημα και πάλι πολύ ευαίσθητο. Είναι η αποστολή των συστάσεων του Όλαφ προς τις κυβερνήσεις. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Ο Όλαφ κάνει την ερευνά του, στέλνει τις συστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τις οικονομικές συστάσεις στα κράτη-μέλη. Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια κράτη-μέλη βλέπουμε ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των ενδεχόμενων ε, περιπτώσεων διαφθοράς. Στις περιπτώσει λοιπόν αυτές ε, οι συστάσει του Όλαφ που επιτέλου ε, ερευνούν μια υπηρεσία, μια κρατική υπηρεσία η οποία κατηγορείται ουσιαστικά για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων, τελικά οι συστάσει στέλνονται στην ίδια κυβέρνηση. Ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα η έρευνα αυτό, ενδεχομένω υπονομεύει πάλι τη δυνατότητα που έχει κάθε κυβέρνηση να κάνει σωστή έρευνα. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες αντιφάσεις. Και τέλος, και θα κλείσω στο σημείο αυτό, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Γκρέσλε ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής ε, του Όλαφ θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις για τα ε, ε, το κενό, την έλλειψη ένωμων μέσων κατά των ερευνών του Όλαφ. Δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση σωστά ένωμα μέσα για αυτούς που βρίσκονται υπό έρευνα, υπό εξέταση από τον Όλαφ και το σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων. Εγώ είμαι υπέρ της ενίσχυσης του Όλαφ και της διαβρύνσης ε, των αρμοδιοτήτων τη, αλλά χωρίς το σωστό σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων δεν γίνεται. Πρώτα θα πρέπει να κοιτάξουμε το σύστημα αυτό και μετά να ενισχύσουμε τον Όλαφ καθε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαραβάμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Ερτίνγκερ. Να ευχαριστήσω και την Εποπτική Επιτροπή ο Όλαφ αποτέλεσε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα τα οποία εξέτασα την περίοδο 2012-2015. Δεν ξέρω αν ήσασταν ήδη εκεί. Ο κύριος Μέλτερ θα θυμάται όμως και από την Επιτροπή τα όσα λέγαμε τότε. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα επιτρέψτε μου. Για να υποστηρίξω και αυτά που είπε και ο κύριος, ο προηγούμενος μιλητής και άλλα και η πρόεδρος. νομικός πόσο η κατάσταση είναι εντελώς ε, απαράδεκτη. Το FBI, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εσωτερικό FBI, δεν έχει σωστό νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει σωστό νομικό πλαίσιο, λοιπόν, όταν, για παράδειγμα, παρακολουθεί τους πολίτες ε, και και κάνει υποκλοπές για παράδειγμα σε πολίτες. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω λοιπόν με τους υπόλοιπους αμιλητές. Θα πρέπει να συστήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Και 883 θα πρέπει να εξεταστεί ε, σε βάθος και με εντελέχεια, προκειμένου τέτοια παραθυράκια να κλείσουν στην ε, αναθεώρηση και σε σχέση με το θέμα αυτό. Οι ερευνητικέ αρμοδιότητες, ε, ναι, να διαβριθούν, μάλιστα δεν λέω, αλλά μόνο και εφόσον υπάρχει σωστή νομική ρύθμιση του Όλαφ. Αυτό προφανώς ε, είναι εκ των Δεν είναι δυνατόν. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να διευρυνθούν οι ερευνητικέ αρμοδιότητε χωρί να κλείσουν πρώτα όλα τα παθηνάκια στον κανονισμό και να καθιερωθεί ένα σωστό νομικό πλαίσιο και μια σωστή, ένα σωστό ε, επίπεδο ευθύνη για όλους. Το σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων λοιπόν του κανονισμού πραγματικά θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Και να ζητήσω από την Εποπτική Επιτροπή να μας πει αν σωστά κατάλαβα όλες οι πληροφορίες ακόμα δεν διατίθονται μάλλον η Επιτροπή η Υποπτική Επιτροπή ακόμα δεν ελαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και αυτό Προφανώ είναι απαραίτητο για να είναι σωστό το πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να το πετύχουμε επιτέλου αυτό. Χρόνια το λέμε. Ακόμα που το έχουμε καταφέρει. Τώρα επιτέλους έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να γυρίσουμε και αυτή τη σελίδα στη λειτουργία του Όλαφ. Και τέλο, τα δικαιώματα των ατόμων που είναι υπό εξέταση. θα ήθελα να παραθέσω μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, ένα μέλος του λεκτικού συνεδρίου που βρίσκεται υπό εξέταση. Αυτά μας λέει ο Όλαφ. Ε, εντάξει, να μην γνωρίζουμε εμείς όλες τις πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι το μέλος, ε, ο κύριος Πίνκστεν, θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει ποιο πράγμα ερευνάται. Αυτό αποτελεί πραγματικά ένα ακραίο παράδειγμα για το ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εντελώ απαράδεκτη και δεν μπορούμε να τη δεχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτά και κλείνοντα, συνοψίζοντα, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα, όπω είπε η κυρία Φαζέντα, ότι η Εποπτική Επιτροπή εξακολουθεί να δραματίζει πάρα πολύ επίκαιρο και σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντειούμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ ε, και τον ε, ε, Επίτροπο για την παρουσίασή του αλλά και βεβαίως την Επιτροπή για τη γνωμοδότησή της. Πολλά υπόθηκαν, κάνατε και μια μακρά δήλωση. Κυρία Πρόεδρε, Νομίζω ότι μιλήσατε πραγματικά εξ ονόματος της ε, Επιτροπής και σίγουρα ε, μιλήσατε και εξ ονόματος ε, της δικιάς μου ομάδας. Είδαμε και είπατε και εσείς ποια είναι τα κύρια προβλήματα. Έχουμε τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι απόλυτα λεπτομερής με διαδικαστικά δικαιώματα κτλ. Και εδώ πρέπει να δούμε ποια θέση θα εξακολουθήσει να έχει όλα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η εφαρμογή των ε, κριτηρίων στη διαδικασία επιλογής ε, των υποθέσεων. Είναι ενδιαφέρον ε, να δει κανείς το παράρτημα της αξιολόγησης, <clears throat> γιατί εκεί βλέπει ότι στα εργαστήρια, ας πούμε, καθίσταται σαφές ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν μάλλον επικριτική στάση όσον αφορά την διαφάνεια και την σαφήνεια των διαδικασιών επιλογής ε, υποθέσεων. Και διαβάζοντας ε, την ε, αξιολόγηση της ίδιας της Επιτροπής, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι ε, υπάρχει διακριτική ε, ευχέρεια ε, αλλά λαμβάνοντας και υπόψη ναι, την έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας των κριτηρίων γιατί τα κριτήρια είναι πάρα πολύ γενικά και μπορεί κανείς ε, να τα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Εάν δούμε λοιπόν τα δύο συνδυαστικά, αναρωτιόμαστε με ποιο τρόπο θα ε, προχωρήσει η ε, διαδικασία και πώς, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει και η Επιτροπή και η Εποπτική Επιτροπή το θέμα αυτό. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα, οι διαδικαστικές, τα διαδικαστικά χέγγια. Στο παράρτημα πάντα βλέπουμε ότι όσον αφορά αυτά τα διαδικαστικά ειχέγγυα, σε γενικές ε, γραμμές ε, οι ενδιαφερόμενοι λένε ότι ε, για αυτές τις δικονομικές εγγύησεις λοιπόν, σε γενικές γραμμές ε, οι ενδιαφερόμενοι ε, απαντούν ότι θεωρούν ότι υπάρχει θέμα δυσαναλογίας. Και εάν δει κανεί και τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί ο προβληματισμός μου γίνεται μεγαλύτερος. Γιατί εδώ αναρωτιέμαι από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα δυσαναλογίας, πώς είναι δυνατόν να ε, ε, προχωρήσουμε με τον ε, ίδιο τρόπο από τη στιγμή που καθίσατε σαφές ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια. Η Εποπτική Επιτροπή είπε διάφορα σήμερα και είπε ότι ε, θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος ε, ε, εκπρόσωπος για, τα, για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή εν πάση περιπτώσει να δημιουργηθεί κατά κάποιο χώρο για κάποιο άτομο το οποίο θα ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αυτά είναι απαραίτητα έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις διαδικασίες σχετικά με, την, με τον Όλαφ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πολύ και τον ε, κύριο Επίτροπο καθώς επίσης και τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής για την ε, τοποθέτηση που ακούσαμε όσον αφορά τη λειτουργία του Όλαφ. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σαφώς σε σχέση με το προκείμενο είναι ε, ο Όλαφ να μπορεί να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικός και όσο γίνεται πιο σωστός στην καταπολέμηση της ε, απάτης και στην ε, προσπάθειά του να προασπιστεί τα δικαιώματα, συγγνώμη, τα συμφέροντα, τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι ο Ισπανός συνάδελφος ε, ε, έθεσε πολύ ξεκάθαρα τα θέματα. Εδώ λέμε τρία πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Κύριε Επίτροπε, θέλουμε καλύτερο συντονισμό και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις αρμοδιότητες κρατών μελών. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσα σαφώς να πω ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία και βλέπουμε και το συζητήσαμε και σήμερα κυρία Πρόεδρε ότι δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα, ε, πολύ σημαντικό, ε, των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο συν ε, απόφασης και ο, ο Όλαφ ακριβώς δεν μπορεί να παρέμβει σε ορισμένες χώρες γιατί υπερέχει το εθνικό δίκαιο. Και νομίζω ότι ο Όλαφ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του. Το δεύτερο, ε, μια μεγαλύτερη αποσαφήνιση ε, των δραστηριοτήτων ε, του Όλαφ και, των, και της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έτσι ώστε να μην υπάρξουν επικαλύψεις και σε αστικές και σε ποινικέ διαδικασίες. Και μην ότι υπάρχει ένα άρθρο του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που προβλέπει ακριβώς μια τέτοια συν συνεργασία. Τρίτον, ε, ε, απαιτείται οπωσδήποτε και αποσαφήνιση των δραστηριοτήτων της ε, Όλαφ σε σχέση με τις δραστηριότητες της Εποπτικής Επιτροπής. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα όρια των αρμοδιοτήτων ένθεν και ένθεν. Ε, έχουν υπάρξει μάλιστα ε, και ε, μνημόνια των νομικών υπηρεσιών, υπομνήματα μάλλον των νομικών υπηρεσιών των τριών οργάνων που ακριβώς καταλήγουν, συγκλίνουν μάλλον σε αυτήν την θέση και θα ήθελα λοιπόν να μας, πει την άποψή τους, να μας πούν την άποψή τους επ' αυτού και ο κύριος Επίτροπος και ο πρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής. Επίσης, εδώ γίνεται λόγος για για τον κανονισμό 883 ε, που θα πρέπει να λάβει στην νέα του μορφή υπόψη όλους αυτούς τους προβληματισμούς αλλά εντωμεταξύ θα αρχίσει να λειτουργεί ε, και να ισχύει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι τα χρονικά όρια θα είναι ταυτόσιμα για, τον για την εφαρμογή ε, της, ε, του τροποποιημένου κανονισμού και του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τελευταίο θέμα, κυρία Πρόεδρε, το θέμα του δημοκρατικού έλεγχου ε, της εποπτείας αλλά και της διακυβέρνησης του Όλαφ. Και εδώ έχω μια πολύ σαφή ερώτηση, κύριε Επιτροπέ. Θα δεχόσαστε ο δημοκρατικός αυτός έλεγχος και η αρμοδιότητα να μετατεθεί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε τούτη την Επιτροπή ε, και όχι στην Εποπτική Επιτροπή, όπως ε, συμβαίνει σε όλες τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Και τα... Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα με κάποιο τρόπο ο δημοκρατικός έλεγχος να ασκείται είτε από τούτη την Επιτροπή είτε γενικώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ ευχαριστώ βεβαίω την Επιτροπή, τον κύριο Επίτροπο, καθώ επίση ε, και την Εποπτική Επιτροπή ε, για τα πολύ ενδιαφέροντα που μα είπαν. επανειλημμένα εμεί, σαν Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού, έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί με ενδιαφέρουν ε, οι απαντήσεις σας, αλλά υπάρχει ένα σημείο το οποίο συνδέεται με το πρόβλημα της ε, πρόσβασης ε, στις πληροφορίες. Αναφέρθηκε επανειλημμένα αυτό, δεν είναι πρόβλημα μόνο του Όλαφ, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο αφορά και όλες τις ε, εθνικές ε, υπηρεσίες οι οποίες ας πούμε πρέπει να διεξάγουν έρευνες όσον αφορά διασυνοριακές ε, απάτες και εδώ έχουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Σας ρωτώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, αυτό το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών είναι κάτι που μας προβληματίζει ιδιαιτέρως. Ορισμένες χώρες ε, δεν συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά τουλάχιστον μια συνεργασία μεταξύ αρμοδίων εθνικών ε, ε, αρχών σε περιπτώσεις που θα πρέπει να έρθει το τραπεζικό απόρριτο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να γίνουν έρευνες σε ιδρύματα κτλ. Δεν θα πρέπει για να καλυφθούν αυτές οι περιπτώσεις να υπάρξει μια πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή να υπάρξει μια σωστή τη ε, ανταλλαγή ε, πληροφοριών, ε, αμοιβαία αρρωγή για δικαστικά ζητήματα κλπ. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των καλών ερευνών, αν θέλουμε πραγματικά να ξεσκεπάσουμε απάτες η Επιτροπή ε, Ελέγχου του ε, Προϋπολογισμού ε, έχει επανειλημμένα θίξει το, το θέμα αυτό και η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει σε ποιο πλαίσιο προτίθεται ή θέλει να εφαρμόσει αυτήν την πολιτική τοποθέτηση έτσι ώστε να ξεκινήσει μια καλή συνεργασία επί τη βάση των διαφορετικών ταμείων γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, οι συνάδελφοι έθιξαν πολλά ε, σημεία τα οποία προσυπογράφω και επί των οποίων θα ήθελα να έχω μια απάντηση. Ευχαριστώ. Άλλους δύο έχω. Ο κύριος Βόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο και την ε, ε, Εποπτική Επιτροπή και τον πρώην συνάδελφο Γιάννη Μιλντερ. Χαίρομαι που σε βλέπω, Γιάννη, ενώπιον μας και πάλι. Ε, Όλαφ ήταν ένα θέμα πάρα πολύ επίμαχο στην Επιτροπή μας, επί σειρά ετών. Είχαμε πολλές έντονες συζητήσεις εδώ και πραγματικά ήταν από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε ποτέ για την Όλαφ ε, και επικοδομητική και όλοι κάναμε προτάσεις για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις κλπ. Η δημιουργία τώρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μας δίνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός όλο και στο μέλλον και να το προσέξουμε. Γι' αυτό κάνουμε και τη συγκεκριμένη συζήτηση και γι' αυτό θέλουμε και εμείς να προτείνουμε κάποιες αλλαγές για το μέλλον. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του Όλαφ στο μέλλον. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε την εγγύηση της απόλυτης ανεξαρτησίας, ότι οι έρευνες γίνονται με σωστό τρόπο, πώς επιλέγονται, πόσο διαρκούν, ε, τι γίνεται με τις υποθέσεις, τι συνέχεια δίνεται. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και από την Εποπτική Επιτροπή. Υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Θα πρέπει αυτό να το λύσουμε διαπαντός. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ίσως με ένα σαφή ορισμό το, ε, ποια ενημέρωση θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Εποπτική Επιτροπή ε, για τις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ιδρυθεί με, και θα στηθεί με σωστό τρόπο χωρίς επικαλύψεις με την Όλαφ και όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά κύριε Επιτροπέ βλέπω να διστάζετε να κάνετε μεγάλες αλλαγές. Προτείνετε μία προσέγγιση σε δύο φάσεις για να τροποποιήσετε ε, τον κανονισμό 883 λίγο το 18 και περισσότερο αργότερα. Για ποιο λόγο και τι θα περιλαμβάνει η πρώτη φάση και τι θα περιλαμβάνει η δεύτερη. Να έχουμε έτσι μια γενική εικόνα αυτά που προτείνεται για να γίνονται οι βελτιώσεις και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του όλου, αφού στο κάτω-κάτω όλοι το ίδιο θέλουμε. Ο συνάδελφος Τάκουλα. Okay, thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρεαλιστική ε, στάση που τηρεί. Ο Επίτροπος κατανοεί, νομίζω, ότι δεν μπορούν να γίνουν παράλληλα πάρα πολλές αλλαγές ε, ταυτόχρονα. Να πω δύο λόγια από την ομάδα της Άλντε. Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρονται διάφορες ε, ελλείψεις και προβλήματα του κανονισμού σε ό,τι αφορά την νομική βάση, το νομικό πλαίσιο, την αποτελεσματική λειτουργία του Όλαφ και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με την Υποπτική Επιτροπή. Όλα αυτά τα στοιχεία προφανώς είναι πολύ σημαντικά και σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, στην παρούσα φάση θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις άλλαγες ε, που θα επηρεάσουν και τη μελλοντική προοπτική, τις συστάσεις που έχουν να κάνουν άμεσα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ξεκινήσει να λειτουργεί το επόμενο έτος και είναι κρίσιμο να είναι σωστή και ομαλή εξ αρχής η συνεργασία του με τον Όλαφ. Και προφανώς θα πρέπει να είναι ταχύες οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Την προηγούμενη φορά ε, γίναν σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβλήθηκε το 2016. Οι διαπραγματεύσει ολοκληρώθηκαν όμως το 2000. Ξεκίνησαν το 2006, ολοκληρώθηκαν οι ε, διαπραγματεύσεις το 2013. Και προφανώς θα πρέπει όλες αυτές οι αλλαγές να γίνουν μέχρι το τέλος της θετίας. Αυτό προφανώς από αυτό θα εξαρτηθεί η αποτελεσματική λειτουργία και της Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό οι αλλαγέ θα πρέπει να είναι τεχνική φύσεω, να επικεντρωθούμε κυρίω στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Όλαφ. Η επόμενη, στην επόμενη θετία να γίνουν οι πιο εκτεταμένε αλλαγέ, αν θέλετε. Ο Επιτροπό, λέει η Πρόεδρο. Πρόεδρε. Βουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Η νομική βάση για τον Όλαφα είναι 4 ετών τότε θέλαμε να, πιο, να πετύχουν πιο πολλά. Αλλά αυτά που περιλαμβάνονται στον κανονισμό τη Όλαφ αποφασίστηκε από το Συμβούλιο και από το Κοινοβουλίο. Σχετικά νωρί έγινε λοιπόν η αξιολόγηση. Τέσσερα χρόνια μόλι αργότερα. Δεν είναι και πολύ συνήθες. Έγινε και μια εξωτερική μελέτη, εξωτερική έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Όλαφ. Όποιος τη θέλει να την ε, δει. Και τώρα αναφέρουμε και εμείς και ο κύριος ε, Μούλτερ από την δική του επιτροπή και προετοιμαζόμαστε για μία ανανέωση. Μία, μία ανανέωση του κανονισμού που έχει μόλις ε, κλείσει τρία, τέσσερα χρόνια. Εσείς αποφασίσατε. Και η έκπληξη ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ δεν το πίστευα. Δεν ε, το πίστευα πριν από ένα χρόνο ότι θα το πετυχαίναμε. Και μετά λοιπόν έγινε ένα breakthrough. Και με την Ιταλία. 20 είναι τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν πλέον. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλουμε να ξεκινήσει τις εργασίες της ε, μέχρι τα τέλη του 2020. Η προπαρασκευαστική λοιπόν ε, εργασία για την ίδρυση, με τους διευθυντές, με την task force, όλα αυτά είναι υποπλήρη εξέλιξη και θα πρέπει λοιπόν να τα ολοκληρώσουμε αυτά σε τρία χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε ρυθμίσει και τα συνεργασία μεταξύ ΟΛΑΦ και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην ε, κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουμε το άρθρο 1,1 που αναφέρει τα της ΟΛΑΦ και του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Αυτό είναι το πρώτο και καλύτερο κεφάλαιο, η σχέση της Όλαφ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ έχω να πω το εξή. Δημιουργήσαμε και ιδρύσαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσει κάποιες αρμοδιότητες σε Όλαφ. Για να μειώσουμε τις αρμοδιότητες του Όλαφ. Τα κράτη-μέλη θέλουν να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να αναλάβει όλα αυτά τα καθήκοντα Αυτό είναι πραγματικά διανόητο. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχώ σε ό,τι αφορά τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό για να μπορεί να έχει δυνατότητα δράση η Όλαφ και να είναι και ένα ελκυστικό τόπο εργασία για καλού ε, νομικού νέου ανθρώπου ε, με κίνητρο. Βέβαια, όπω τα δείκανε στα τα πράγματα, μισογεμάτα ή μισοάδια, τουλάχιστον μισογεμάτο. Έχω καλή εντύπωση για την όλα Να σας πω την αλήθεια. Πολύ καλή εντύπωση. Έχω μιλήσει με διάφορα άτομα που εργάζονται και είναι πραγματικά και ικανά και έχουν και στη σωστή στάση. Έχουμε ένα εξαιρετικό διευθυντή και ε, είμαι ευγνώμων προς τη γυναίκα του που τον έπεισε να λάβει αυτά τα καθήκοντα. Είμαστε σε στενή επαφή και θα Υποβάλλουμε ένα κατάλογο ε, υποψηφίων ε, στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Έχουμε λοιπόν ήδη ένα κατάλογο με υποψηφίους προκειμένου την άνοιξη να αναλάβει τα καθήκοντά του ο ή η διάδοχος του διευθυντή. Εδώ και χρόνια ήταν ε, α, μόνιμος αντικαταστάτης του διοικητή. Παρακαλώ λοιπόν να δεχτούμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι χρειάζεται από νομικής άποψης και μόνο σε περιορισμένο βαθμό αυτό που θα θέλατε από πολιτικής άποψης να συμβεί. Γνωρίζω τον κανονισμό της Όλαφ ε, και είμαι βέβαιος ότι και εγώ και η Όλαφ επιτελούμε όλα μας τα καθήκοντα. Αναφέρθηκε το θέμα του ελέγχου. Πολύ σωστά. Υπάρχει και κάναμε πρόταση για τριετή έλεγχο. Δικαίως το παγώσατε αυτό ως πρόταση, προκειμένου να γίνει πρώτα η αξιολόγηση της Όλαφ. Τώρα όμως μπορούμε αυτό το θέμα να το κοιτάξουμε από κοινού γιατί υπάρχουν και εν μέρη ζητήματα τα οποία μπορούμε ασφαλώς να τα συζητήσουμε, αλλά ο έλεγχος ήταν καθεαυτός πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε η περίπτωση έρευνας ενός ε, ε, μέλους Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου. Σας παρακαλώ προσοχή γιατί εδώ πέρα έχουμε εμπιστευτικό χαρακτήρα, πιο προραίο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Και η υποχρέωση μιας, υποχρε... μιας ε, υπηρεσίας όπως η Όλαφ ε, να τηρεί απόρριτο σε ό,τι αφορά τα ονόματα και τις διαδικασίες και τις έρευνες για οποιοδήποτε άτομο. Μιλάμε για κράτο δικαίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στην Όλαφ δεν τηρείται το τραπεζικό απόρριτο ε, και δεν ε, τηρούνται οι... και δεν τηρούνται τόσο θα πρέπει να τηρούνται από πλευρά εμπιστευτικότητα και παράλληλα να μιλάτε για νόματα εδώ πέρα. Χωρίς εμπιστευτικότητα η Όλαφ είναι μια υπηρεσία που κάνει διοικητικέ έρευνε. Δεν συγκρίνεται με το FBI. Το FBI από τη δομή του και από τα καθήκοντα τα οποία έχει και φυσικά και από το βαθμό που είναι γνωστός στον κόσμο, ε, κάτι τελείω διαφορετικό. Οι, οι υπάλληλοι της Όλαφ δεν έχουν ρεβόλβερ. Πώς να το κάνουμε. Έχουν μόνο την εμπειρογνωμοσύνη του το θέμα των κρατών μελών και της πρόσβασης και της διαφάνειας το αναφέρατε. Εμείς όλοι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Και είμαστε από ένα κρατός μέλος, όλοι μας. Εγώ από τη Γερμανία, από την Ουγγαρία, από την Ιταλία, από την Ελλάδα, ο καθένας από τη χώρα του. Δυστυχώς, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η Ευρώπη των εθνικών κρατών μελών. Άρα είναι ισχυρό το Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πλήρεις ε, αρμοδιότητες ε, νομοθετικές ε, στα χέρια του Κοινοβουλίου. Προς τα κοιοδεύουμε Αλλά οι εθνικοί οι υπουργοί, οι τοπικοί υπουργοί, οι τοπικές έτσι, κυβερνήσεις θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, αν θέλετε, ο προϊστάμενος τους. Και άρα το θέμα της διοικητικών αρμοδιοτήτων και των πενικών διώξεων θεωρείται εξοχήν εθνική υπόθεση, εθνική αρμοδιότητα. Από το Ελσίνκι, από το Βερολίνο, μπορούμε να καθόμαστε όλοι μαζί, να πίνουμε και ένα πιτρικασί και να λέμε ναι, ναι, ναι, διαφάνεια, πλήρης πρόσβαση. Μπορούμε να το βάλουμε και να το κάνουμε. Αλλά όσο δεν το καταφέρουμε να το κάνουμε στη Ρώμη, στην Αθήνα, στη Βουδαπέστη, στο Βερολίνο, Α είμαστε τουλάχιστον ρεαλιστέ στην καριέρα μα την υπόλοιπη. Ε, εξηγήσαμε το τι θέλουμε να προτείνουμε και σας είπα ότι θα συμπεριλάβω και κάποιες από τις προτάσεις για την Υποπτική Επιτροπή και θέλω πριν το Μάρτιο να κάνουμε συζητήσεις με τον κύριο Μίλντερ και τα μέλη της Επιτροπής του. Αλλά θα ήθελα να γίνει και ένα, μια ψηφοφορία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Συγγελία ξεκινάει το 2020. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί νομοθεσία για τον Όλαφ. Και από τριμερίου διαλόγου γνωρίζετε τι γίνεται στο Συμβούλιο. Ξέρετε πώ έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Πιστεύετε πραγματικά δηλαδή ότι αν ε, εκφράσω όλες τις σκέψεις από πλευρά σας και τις βάλω σε ένα πακέτο. Είναι σοβαρές, δεν λέω. Πιστεύετε ότι το πακέτο αυτό θα έχει περάσει μέχρι το Μάιο του 2019. Με καμία δύναμη. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε πάρα πολλή εμπειρία στην νομοθετική διαδικασία για να μην το πιστεύετε αυτό. Τέσσερα χρόνια χρειαστήκαμε για την Ευρωπαϊκή Συγγελία. Ε, περισσότερα πέντε χρόνια χρειάστηκε το, το Γι' αυτό λοιπόν στην υπόλοιπη θετία σας ας κάνουμε μια σωστή διάκριση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Αγγελίας και Όλαφ. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ΦΠΑ και τον Όλαφ. Αν θέλετε να το κοιτάξουμε αυτό θα το κάνω, αλλά να το κάνουμε σε ένα σωστό ε, πακέτο. Και τότε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο, προκειμένου το Συμβούλιο, η Βουλγαρική Προεδρία συγκεκριμένα, η Αυστριακή και η Ρουμανική Προεδρία να τα έχουν ολοκληρώσει αυτά, να τα έχουν αποφασίσει μέχρι Απρίλιο-Μάιο του 2019. Και τότε, χωρίς χρονική πίεση, ας κάνουμε έναν ενδελεχή, μια ενδελεχή αναθεώρηση και α συμπεριληφθούν όλες οι ανησυχίε και οι σκέψεις σας σε ένα δεύτερο συνεκτικό πακέτο. Τουλάχιστον όμως μέχρι τότε να λειτουργεί σωστά η Όλαφ. Σωστά είναι τα θέματα που σας απασχολούν. Εμένα αυτό που με απασχολούν είναι η ταχύτητα και φυσικά περιορισμένα στοιχεία. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν αποτελεί αντίφαση Εξορισμό. Στο πρόγραμμα εργασίας 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο και γνωρίζετε, το οποίο ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο, ακριβώς αυτή την προσέγγιση ε, αναφέραμε. Σας είναι γνωστά όλα αυτά. Αν θα θέλαμε μια ευρύτερη προσέγγιση, θα πρέπει να κάναμε διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων υποχρεωτικά. Και θα έπρεπε υποχρεωτικά να κάνω μελέτη δικτύπου. Η δική μου πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή είναι ότι το νωρίτερο στα τέλη του 2018 θα τα πετυχαίναμε αυτά. πριν από την, εργασία, από την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ε, δεν θα έμενε χρόνος όμως. Ε, θα είχαμε μόνο δηλαδή μέχρι τότε ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο θα χρειαζόταν ε, να το κοιτάξει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο ξέρει τι θα το έκανε. Κάποιοι εξημών θα συμμετέχετε και στο επόμενο κοινοβούλιο, κάποιοι άλλοι όχι αλλά η εμπειρογνωμοσύνη σας είναι σημαντική. Ας ασκήσουμε πίεση λοιπόν με αυτή την εμπειρογνωμοσύνη σας στο Συμβούλιο προκειμένου να καταθέσει μια πρόταση ε, μεταρρύθμισης ε, μέσα σε ένα χρόνο να την ψηφίσει αυτή την πρόταση. Ένα πρώτο τελευταίο σημείο, επιτρέψτε μου. Η βασική μου ανησυχία είναι το σχέδιο το της Όλαφ, του Όλαφ, γιατί και ο Όλαφ έκανε περικοπές 5%. Αυτό που με απασχολεί λοιπόν είναι να υπάρχει επαρκή αριθμό ε, ικανών υπαλλήλων. Έχουμε αρκετέ θέσει. Είμαστε ω εργοδότη ε, ελκυστικό. Υπάρχουν δυνατότητε σταδιοδρομία ε, στην Όλαφ. Είμαστε ελκυστικοί ω εργοδότε. Και Θα ήθελα τα επόμενα στο τίτλο 5 να προσθεθούν ε, θέσεις ε, στην όλα αυτά τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και ούτε εσείς είστε ικανοποιημένοι με την φυστάμενη κατάσταση. Είναι τα προγράμματα όπως είναι και δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, οποιαδήποτε υποδομή για τέτοια ζητήματα οι αρχές μας για τα μεικτά προγράμματα, οι υπηρεσίες μας για τις ε, περίπλοκες ε, ευρωπαϊκές νομοθεσίες είναι οι δήμοι, οι κοινότητες, οι εθνικές ε, αρχές και δυστυχώς είναι όπως έχουν. Άλλοι είναι καλύτεροι, άλλοι λιγότερο. Δεν έχουμε άλλους όμως. Έχουμε 28 κράτη-μέλη, 200 περιφέρειες, χιλιάδες δήμους και κοινότητες. Αυτή είναι η κατάσταση. είναι σε μερικέ περιπτώσει εξαιρετικέ οι αρμοδιότητε διοικητικέ, σε κάποιε άλλε όμω όχι. Αλλά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ήπειρο ε, τη διαφθοράς και ξέρω πάρα πολλούς δημόσιους υπαλλήλους σε πάρα πολλά επίπεδα συμμετείχα ε, στη δημόσια διοίκηση χιλιάδες υπαλλήλους της Κομισιόν γνωρίζω η μεγαλύτερη συντριπτική πλειοψηφία έχει σωστή στάση είναι εμπιστευτική ε, αξίζει την εμπιστοσύνη μας και είναι πάρα πολύ ικανή και δεν θέλει να προαγάγει την διαφθορά δεν θέλει να υπάρχει καν διαφθορά φυσικά δεν ε, ξεφάβουν κάθε περίπτωση διαφθοράς αλλά νομίζω ότι η φε έχει πραγματικά πολύ σωστή και αποτρεπτική δράση. Γιατί όταν παίρνουμε καταγγελίες για ε, κατηγορίες ε, διαφθοράς, τις εξετάζουμε. Και έτσι δρά αποτρεπτικά η Όλαφ. Το τελευταίο είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Μισογεμάτο, όχι μισοάδιο το ποτήρι. Και η Όλαφ είναι μια υπηρεσία η οποία αξίζει την εμπιστοσύνη μας, την έχει κερδίσει. Και ο Γενικός Διευθυντής με την εμπειρία του όλο ιδιαίτερος. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου ο νέος ή η νέα Γενικός Διευθυντής, Γενική Διευθυντρία να είναι κάποιος που θα εγκρίνεται και που θα εγκρίνει και η Υποπτική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, αλλά ξέρετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας απασχολεί ο Όλαφ. Και ε, το να ωρεοποιούμε την κατάσταση ευτυχώς δεν μας ικανοποιεί πλέον. Τα έχουμε ξανακούσει. Τα προβλήματα που έχουμε πρέπει να τα λύσουμε. Και όχι να προσπαθούμε πάντα με κάποιο τρόπο να τα παρουσιάζουμε και να μην τα αναβάλουμε τώρα επαόριστα, να τα λύσουμε επιτέλους. Και θα κάνουμε και τροπολογίες, 120 την περασμένη φορά, τώρα δεν ξέρω κάποιες εκατοντάδες. Ήταν πάρα πολύ επίπονη η διαδικασία με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φτύσαμε αίμα γενικώ με όλους τους ενεχομένους. Εμένα μου αρέσει αυτό το εγχείρημα και χαίρομαι. Αλλά δεν βοηθάει πια να μένουμε στα λόγια. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να αποσύρει τον έλεγχο μετά από δική μας παράκληση. Ε, είπαμε να μην βγει. Ε, το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται. Ε, πάντως τώρα μου μπαίνει και όρεξη να το κάνω, να δούμε ποια είναι η άσκηση στην οποία θα επιδοθούμε για να αποκρισταλώσουμε θέση. Βεβαίως, είναι σε πλήρη συναπόφαση ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή και κανονικά θα ήταν στην στην απόφαση και ο ασκών καθήκοντα. Από το 2011 είχαμε εκτενή αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό έχουμε εξασκηθεί. Αλλά σύντομα τελειώνουμε. Να μην συνεχιστεί αυτή η παλιά αλληλογραφία. Τα ε, θέματα είναι γνωστά και οι θέσεις είναι γνωστές. Άρα θεωρούμε ότι ο Γενικός Διευθυντής ή αυτός που ασκεί ε, καθήκοντα ε, διοικητού μας, μας αφορά και μας και θα έπρεπε να έχουμε λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Μόλτερ και μετά η κυρία Φαζέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, κάνατε κάποιες σημαντικές ε, παρατηρήσεις για ενδεχομένες αλλαγές στην οδηγία. Με χαρά να το συζητήσουμε μαζί σας, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αναφέρετε και πρέπει να λυθούν. Συμφωνώ. Και αυτό φορά και τον Επίτροπο. Είμαστε απολύτω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρώτον, τα σχόλια που έκανε ο κύριος Γιάβορ και ο κύριος Σάβαρμα. Συμφωνούμε απολύτως είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφέρον της όλα να λειτουργεί σωστά με αντίβαρα και με ελέγχους. Θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί στο έργο μας, να μην ε, προβάλλουμε άχρηστες δυσκολίες και περιτές, αλλά είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα να είναι ανεξάρτητο όργανο και ένα ανεξάρτητο επίσης εποπτικό όργανο να τα ελέγχει όλα αυτά και χρειαζόμαστε την ενημέρωση, την πληροφόρηση ε, γι' αυτό. Είχαμε διάφορες προφάσεις στο παρελθόν για το αντίθετο και για να μην γίνει παρεξήγηση δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο του Γενικού Διευθυντού. Θα πρέπει να αναφέρεται στην νομοθεσία ότι θα πρέπει κάποια ελάχιστη πληροφόρηση να έχουμε και στην Εποπτική Επιτροπή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ποια θα είναι αυτή η πληροφόρηση, θα το συζητήσουμε. Διαβάζοντα όμως τις αιτήσεις εκθέσεις των τελευταίων ετών, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε χρόνο λέμε ότι δεν πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και πάλι, αν είμαστε ανεξάρτητοι και οι δύο επιτροπές και, και η Επιτροπή μας και η Όλαφ, αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με τον κύριο Ντι ότι χρειάζονται σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση. Μα γι' αυτό άλλωστε το λέμε και στη δική μας έκθεση. Δεν αρκεί να δημοσιεύονται κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να είναι και τμήμα της νομοθεσίας. Ε, αυτό εξαρτάται βέβαια από τον νομοθέτη για να είναι ε, σαφής οι ενδείξεις διαφανής, ε, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει όλα. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση θα το ψάξω, είναι καινούριο αυτό που μου λέτε, θα το κοιτάξω. Περίεργο μου φαίνεται πάντως. Προφανώς όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια είτε είναι στη συνυπευθυνότητα, είτε είναι στην 100% ε, χρηματοδότηση, παραμένουν ευρωπαϊκά κονδύλια και θα, μπορεί, θα πρέπει να μπορεί Μαρόνι όλα αυτά να το διαρευνά. Θα το κοιτάξω, δεν έχω σήμερα να σας δώσω σαφή απάντηση και ακριβή. Ο κύριος Βάλη τώρα αποχώρησε. Κύριε Βόν, νομίζω απάντησα πάνω κάτω σε αυτά που ρωτήσατε η Ελένα Φαζέντα, φυσικά με την άδεια της Προέδρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Με εξαίρεση τις γενικές παρατηρήσεις που έκανε μόλις ο κύριος Μόλντερ. Πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε γιατί πολλοί βουλευτές κατέδειξαν τις δυσκολίες που υπάρχουν με την Όλαφ και με την Εποπτική Επιτροπή. Ρώτησαν πολλά οι ε, βουλευτές με πολλές λεπτομέρειες. Εμείς προσπαθούμε πάντα να είμαστε επικοδομητικοί και να συνεργαζόμαστε μαζί σας και πάντα στη διάθεσή σας. Και κάθε φορά που παίρνουμε το λόγο είναι παρόν και ο Γενικός Διευθυντής όταν δραστηριοποιείται η υπηρεσία Όλαφ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πραγματικό προνόμιο ευκαιρία όσο και δυνατότητα να ορίσουμε τώρα ακριβώς για τον Όλαφ σε ένα κανονισμό ποιες είναι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του. Πότε μπορεί να κάνει έρευνες, με ποιες πρακτικές, όλα πάρα πολύ συγκεκριμένα και περιγεγραμμένα. Αυτό θα κάνει το συγκεκριμένο όργανο ακόμα πιο αποτελεσματικό στη λειτουργία του όταν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την απάτη, τη διαφθορά και άλλες παρατυπίες και ατασταλίες. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το θέμα, διότι ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνει ήδη ρητή αναφορά για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί. Παραμένουν κάποιες διευκρινήσεις μόνο Και υπάρχουν κανόνες σε δύο επίπεδα. Πρώτον, κανόνες για τη δεξαγωγή της έρευνας. Τι θα πρέπει να κάνουν οι διάφοροι αρμόδιοι για την έρευνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι θα επιτρέπεται και τι θα απαγορεύεται. Βεβαίως με δικονομικές εγγύησεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα να παραμένουν εξασφαλισμένα. Εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία αυτή που θα πρέπει να βρεθεί. Και φυσικά όλα αυτά τα χρόνια ο Όλαφ κατάφερε να βελτιώσει τη λειτουργία και τις έρευνες, αλλά πάντα καλύτερο είναι να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Θα πρέπει να είναι σωστή η εσωτερική δομή του Όλαφ. Όπως κάνουν όλα τα διοκτικά όργανα ή τα εξεταστικά όργανα, υπάρχουν ε, καθορισμένοι, προκαθορισμένοι τομείς αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις ικανότητες και τα καθήκοντα. Ποια μονάδα κάνει ποια έρευνα, ποια μονάδα στην Όλαφ ασχολείται με συγκεκριμένα αδικήματα πώς γίνεται η ανταλλαγή των στοιχείων και των πληροφοριών στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Όλαφ. Αυτό θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα των ερευνών, γιατί ταυτόχρονα έχουμε κανόνες λειτουργίες, κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών και διαβίβαση πληροφόρησης στην Υποπτική Επιτροπή για να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει ένα μνημόνιο της συνεννόησης από το 1999 για το πώς διαβιβάζονται αυτές οι πληροφορίες στην Εποπτική Επιτροπή. Και ουσιαστικά δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα ποτέ. Ο κανονισμός υπάρχει, βελτίωση φυσικά χωράει πάντα και τελειοποίηση ακόμα περισσότερο. και θα πρέπει να γνωρίζει όλα τι μπορεί και τι οφείλει να διαβεβάζει στην Επιτροπή μας. Η δική μας Επιτροπή είναι ένα όργανο ανεξάρτητο με εγγυήσει για την υποπτία της λειτουργίας ε, της υπηρεσίας αυτή. Και από τα τρία θεσμικά όργανα έχουμε διοριστεί και εκεί δράζεται και η εντολή μας. Είμαστε λοιπόν πάντα πρόθυμοι να συνεργαζόμαστε και να σας διαβάζουμε τις προφορίες που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το θέμα στην μέση διάταξη. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη όλοι για το θέμα του διοργανικού διαλόγου. Σας ευχαριστούμε και δεν θα χαθούμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Πίτροπε, και Διευθυντά. Μπορείτε να παραμείνετε κύριε Άλπ. Συνέχιση της παρακολούθησης της αιτήσιας έκθεσης του 2016 για την πρόσβαση στα έγγραφα, να δούμε τι έχει γίνει. Παρακαλώ, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την πρόσβαση στα έγγραφα. Uh, until now... Ναι, κυρία Πρόεδρε. Μέχρι τώρα κοίταξα, μελέτησα διάφορα προβλήματα τα οποία είχαμε και στο παρελθόν και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση με την ε, Όλαφ και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία είναι θετική. Προσδοκούμε ε, ε, καλή συνεργασία. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ε, για να πούμε ότι τα πάντα είναι εξαιρετικά, αλλά πάντως εμφανίζονται αρκετά θετικά. ακούω και τις επικρίσεις του όλα. όσον αφορά την ετήσια έκθεση της ε, Εποπτικής Επιτροπής για το 2016. Εμείς μπορούμε να απαντήσουμε εν λεπτομερία σε όλα τα σημεία Έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν προετοιμάσαμε την ε, ε, ε, έκθεση της φετινής χρονιάς ε, ελπίζουμε, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη αρχή της επόμενης χρονιάς, ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα ε, να έρθουμε σε επαφή με τον Όλαφ, δηλαδή να έχει ο Όλαφ την δυνατότητα να σχολιάσει πριν δημοσιευθεί το περιεχόμενο Ε, γιατί την προηγούμενη χρονιά η δημοσίευση έγινε το Μάιο και ο Όλαφ έκανε τα σχόλια και τις επικρίσεις τον Ιούλιο. Οι επικρίσεις ε, αφορούν ε, το θέμα της δυσκολίας όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον μπορεί να αποφασίσει η Όλαφ σε ποιες περιπτώσεις για τις οποίες έχουμε ήδη αιτηθεί πληροφορίες ε, θα δώσει συνέχεια ή όχι. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι ε, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει την επιλογή. Πάντως η μεγαλύτερη διάσταση απόψεων στο παρελθόν αφορούσε το θέμα αυτό. Πάντως ευελπιστούμε ότι ε, μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία και σε ορισμένους ε, μήνες ίσως να είμαι και σε θέση να σας πω ακριβώς ποιε είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τα θέματα αυτά. Πάντως τα πρώτα μηνύματα είναι μάλλον θετικά και είμαι μάλλον αισιόδοξο. Εάν θέλετε τώρα θα περάσω στα επόμενα σημεία, συγκαταλέγετε θετικά, οπότε συνεχίζω. Η έκθεση είναι έκθεση της προηγούμενης ε, επιτροπής και όχι της ε, ε, τωρινής αυτής της επιτροπής του 2016 αλλά αυτό είναι μια επίκριση του Όλαφ αλλά εμείς αποτελούμε συνέχεια της προηγούμενης επιτροπής επομένως και η άσκηση αυτής της δραστηριότητας αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας και επομένως υπεραμεινόμεθα του περιεχομένου αυτής της εκθέσεως. Υπάρχει και ένα άλλο ε, ερώτημα. Γιατί η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες μονάχα για μία υπόθεση το 2016 για πρόσβαση στα ε, στοιχεία και δεν ικανοποιήθηκαν με τις ε, πληροφορίες που πήραν. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ζητήσει πληροφορίες για διάφορες υποθέσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν ε, ελήφθησαν ικανοποιητικές αποτελέσεις. Τώρα, πέρσι μπορεί να ζητήθηκαν πληροφορίες για μία μονάχα υπόθεση στη Γαλλία, αν ε, δεν κάνω λάθος. Αλλά η απάντηση δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Και επομένως, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και το σημείο αυτό. Το ερώτημα είναι γιατί η Επιτροπή δεν δέχτηκε, αυτή η ε, Επιτροπή δεν δέχτηκε ε, τις ε, προτάσεις του Όλαφ. Κοιτάξτε, όταν διερευνά κανείς κάτι, θες να το κάνεις με τους δικούς σου Θες, να κάνεις την έρευνα μόνο σου και εντάξει αυτό μπορεί να είναι λογικό αλλά ερώτηση. Γιατί η πρόσβαση στις 62 υποθέσεις που αφορούν την διάρκεια των ερευνών αναφέρεται μονάχα σε υποσημείωση σε μία και μόνη σελίδα. Τώρα, είτε βρίσκεται σε υποσημείωση ή όχι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Κατά την άποψή μας, το γεγονός ότι βρίσκεται σε υποσημείωση δεν ε, μειώνει τη σημασία της αναφοράς. Κοιτάξτε, τι δηλαδή, δεν ξέρω δεν νομίζω ότι ε, είναι τόσο σημαντικό. Ε, τώρα, εάν ε, ο Όλαφ προσβλήθηκε από την αναφορά σε αυτήν την υποσημείωση, εντάξει, θα το διορθώσουμε ενδεχομένως. Μπορούμε να τα συζητάμε αυτά από καιρούς καιρών. Κάποιες συστάσεις για ευαίσθητες υποθέσεις, εάν δεν απαντηθούν από τον Όλαφ, που δεν έχουν μάλλον απαντηθεί από τον Όλαφ. Αλλά εδώ υπεύθυνο ε, δεν είναι ο Όλαφ, αλλά η Κομισιόν, ε, η οποία δεν έδωσε τις απαραίτητες ε, πληροφορίες. Το επίπεδο είναι διαφορετικό. Ίσως θα έπρεπε αυτό να το έχουμε αναφέρει στην έκθεση πιο ξεκάθαρα. Τέλ, επίσης. Η διάρκεια των ερευνών. Αυτό μας προβληματίζει αναφέρεται και στην έκθεση άλλωστε. Όλαφ λέει, σας δώσαμε τόσα έγγραφα, Και τώρα εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε νέο διάλογο πάντως με τον Όλαφ για την ε, διάρκεια. Γιατί με πολύ μεγάλη τσιγκουνιά και, και, και φιδωλά έτσι μας δίνουν ε, τις ε, πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Και θα δείτε ότι σε πολλές περιπτώσεις το Google να το αναφέρεται ότι η τάδε ή η η δίνε υπόθεση δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω ελλείψεως ε, σωστής πληροφόρησης. Την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε και έναν μακρύ κατάλογο ε, με υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ε, ολοκληρωθεί και επομένως θα ακολουθήσουμε την πρότασή σας. Ε, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε το, την αιτία της καθυστέρησης. Ωστόσο υπάρχει κάποια πρόοδος και νομίζω ότι αυτό θα το αναφέρουμε στην επόμενη έκθεση αξιολόγησης. Ε, οι ρυθμίσεις εργασίας. Ε, η Επιπτική Επιτροπή ε, είπε ότι δεν χρειάζονται working arrangements. Με την έννοια ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν ήταν απαραίτητες μετά από τα υπομνήματα των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων. Εκεί ρητά αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία είναι αποδεκτά και αυτά τα οποία δεν είναι αποδεκτά. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απολύτως με την τοποθέτηση των νομικών ε, υπηρεσιών. Και επίσης και ο κανονισμός του άρθρου του 3 είναι πάρα πολύ σαφής και ρητά αναφέρει. Και ο κανονισμός 883 ε, είναι σαφής όσον αφορά τα θέματα αυτά. Όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Όλαφ ε, σταμάτησε ε, αυτές ε, τις ρυθμίσεις εργασίας, αλλά λυπάται που το έκανε, μετάνιωσε. Είχαμε μια συνάντηση και ε, ζητήσαμε να, να ξαναδούμε την κατάσταση, ε, να δούμε εάν αυτά τα working arrangements μπορούν ε, να λειτουργήσουν, εάν όμως γίνουν με καλύτερο τρόπο. εάν δεν υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση των ε, στην πρόσβαση στις ε, πληροφορίες. Ε, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια λύση. Σε αντίθετη περίπτωση όμως θα αντιταχθούμε. Θα πρέπει να, να βρεθεί κάποια λύση για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά στο παρελθόν και θα πρέπει να το ξαναδούμε. Και ε, το ίδιο ισχύει ε, και με τα παράπονα τα οποία φτάνουν ε, στον Όλαφ. Η Εποπτική Επιτροπή δεν έχει αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία αυτά. Τώρα αναφέρομαι για την έκθεση. Όσον αφορά τώρα τα στατιστικά στοιχεία, Όλα αυτά ε, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος που σε καθημερινή περίπου βάση ε, ασχολείται με τα στοιχεία αυτά. Αλλά φαίνεται ότι και αυτά η Όλαφ δεν τα έχει δεχτεί ε, με ικανοποίηση, αλλά είπα και προηγουμένως ότι θα στείλουμε την επόμενη ετήσια έκθεση ε, έγκαιρα και πρώτα στον Όλαφ, έτσι ώστε να τον, την μελετήσει και να κάνει τα σχόλιά του. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σαφής όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, παρακαλώ πολύ να μας ε, υποβάλλετε τα σχόλιά σας και βεβαίως ε, ε, θα το δούμε αν πρέπει να αλλάξει κάτι γιατί οτιδήποτε δημοσιεύεται θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους και αν ο ίδιος ο Όλαφ δεν έχει ξεκαθαρισμένη άποψη σχετικά με τα στοιχεία τότε σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Επίσης η διάρκεια των ερευνών είναι υπερβολική θα πρέπει και αυτό να βελτιωθεί. Στη συνέχεια, ε, πειθαρχικές συστάσεις. Θα θέλαμε να είμαστε πιο ενημερωμένοι ε, από ότι είμαστε στην παρούσα φάση. Για τη δειγματοληψία τώρα των ε, υποθέσεων θα πρέπει να κάνουμε συμφωνίες, να κάνουμε κάποιες συμφωνίες γιατί αυτό δεν επαφίεται και πάλι μόνο στον Όλαφ. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή συμφωνία από αυτού. Και τελευταίο στοιχείο. Η Επιτροπή έλαβε πάνω από 800 σελίδες πληροφορίες για τις δικαστικές συστάσεις στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 850 σελίδες αποτελούν ε, μεγάλο όγκο πληροφοριών και ο αριθμός των σελίδων, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στον όγκο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα. Τι πληροφορίες είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για μας. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Ούτε αυτό ήταν ε, σαφές. Ε, και ελπίζω ότι με αυτά, Πρόεδρε, αν και δεν είμαι βέβαιος, Ελπίζω να απάντησα πιο, τα πιο πολλά ερωτήματα της Επιτροπής ΟΛΑΦ ε, ε, και παρακαλώ μην διστάσετε να μας θέσετε ερωτήσεις. Αν το επιθυμείτε θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Σε κάποιες περιπτώσεις ούτε και εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σκεφτώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, τοποθέτηση αυτή. Να δώσω το λόγο και στην Όλαφ να πάρει το λόγο για να μιλήσει. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε και είναι τιμή και προνόμιό μας να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Δεν το περίμενα. Τώρα κατά πόσον θα είναι χαρά μας δεν ξέρω. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον πρόεδρο της Εποπτικής Επιτροπής για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Το πρώτο σημείο που ήθελα να θίξω είναι το εξή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά των τελευταίων ετών. Νομίζω ότι ο διάλογο διακατεχόταν από έλλειψη επικοινωνία, πραγματική επικοινωνία τα τελευταία χρόνια, σε όλα τα επίπεδα μάλιστα, όχι μόνο μεταξύ των ε, επικεφαλής, αλλά πραγματικά σε όλα τα επίπεδα υπήρχε έλλειψη επικοινωνία. Από πλευρά μου είμαστε και ο πρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι και αποφασισμένοι να το διορθώσουμε αυτό και να γίνει μια σωστή συζήτηση για τα θέματα που ανακύπτουν σήμερα και που ανακύπτουν αν θέλετε και στην έκθεσή σας γιατί από πολλές απόψεις θα μπορούσαμε να τα επιλύσουμε τα θέματα αυτά αν συζητούσαμε καλύτερα και καλωσορίζω ιδιαίτερως ε, την απόφασή σας να μοιραστείτε το σχέδιο της επόμενης ετήσιας έκθεσης προκειμένου να απαλείψουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση και μου είπαν ότι σε πολλές περιπτώσεις το παρελθόν ναι, χορηγήσαμε ή εν πάση περιπτώσει προσφέραμε κάποιες πληροφορίες. Θεωρήσαμε ότι είχαν ε, διαβιβαστεί αυτές οι πληροφορίες και δεν ε, λάβαμε απαντήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές που είχαμε αποστείλει. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε αυτό σε, σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες εδώ στην Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, για να μην σας ε, ε καθυστερούμε. Αλλά αυτό σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί στο μέλλον. Ε, η συζήτηση που ε, είχε η Επιτροπή σας στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξετάσατε τι είδους αλλαγές θα ήταν ευκτές και απαραίτητες. Στην παρούσα φάση λειτουργούμε σε ένα νομικό πλαίσιο που ζητά από την Επιτροπή να ζητά πληροφορίες και να αιτιολογεί τις πληροφορίες αυτές που ζητά. Ιδάλλως δεν μπορούμε να χορηγήσουμε τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, χορηγούμε τις πληροφορίες αυτές όποτε το μπορούμε. Όποτε μπορούμε. Έχω δώσει μεγάλη πρόσβαση σε στοιχεία τις τελευταίες εβδομάδες. Στοιχεία που έχουν ζητήσει, που έχει ζητήσει η Υποπτική Επιτροπή. Κάποιες ε, από αυτές τις πληροφορίες ε, είναι πολύ ευαίσθητες. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Και προσπαθούμε επίσης στην παρούσα φάση να επιλύσουμε διάφορες τεχνικές δυσκολίες που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Και μιας και το έχετε ήδη ζητήσει στο προηγούμενο σημείο της Μερικής διάταξης, θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι εδώ και χρόνια έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για την ε, βελτίωση των βασικών ε, συστημάτων IT, τα συστήματα OCM όπως ονομάζονται. Αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε πολύ παραπάνω πράγματα από αυτά που κάνουμε στην παρούσα φάση. Και να αντικαταστήσουμε και ένα σύστημα το οποίο ήταν τεχνικώς παροχημένο και δεν μπορούσε πλέον να συντηρηθεί επαόριστον. Αναπτύσσουμε λοιπόν το σύστημα αυτό μόνοι μας με την χρήση και εξωτερικών ε, εμπειρογνωμόνων υπό την άμεση καθοδήγησή μας, αλλά αντιμετωπίζουμε πιο μεγάλα προβλήματα από ό,τι αναμενόταν. Αυτό προφανώς αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα και δεν είναι και κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα συστήματα IT. Τέτοια προβλήματα τακτικά παρουσιάζονται. Βασική μου λοιπόν προτεραιότητα είναι να τα επιλύσουμε αυτά το συντομότερο δυνατόν πρωτού τουριστεί ο επόμενο Γενικό Διευθυντή. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω είναι το εξή. Παρά το γεγονό ότι το σύστημα παρέμβαση για πρόσβαση σε μεμονωμένα έγγραφα είναι κάτι το απαραίτητο, υπάρχει πλήρης, μητρό όλων αυτών στο σύστημα. Άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνο σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα του οποιοδήποτε εγγράφου, οποιαδήποτε αίτημα έχει κατατεθεί έχει καταγραφεί και ο ετών για τις καταγγελίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χορηγούμε στην Επιτροπή καταλόγους με τις καταγγελίες που έχουμε λάβει καταγγελίες που έχουν γίνει και από άλλες αρχές ε, και έχουν γίνει και προς άλλες αρχές, προς το δικαστήριο, προς τον διαμεσολαβητή. Δεν είναι πολλά, ξέρετε. Δεν είναι πολλές αυτές οι υποθέσεις, πολύ λιγότερες από ό,τι θα φανταζόσασταν σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και προφανώς θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, για τη δειγματοληψία προφανώς δεν ε, αξίζει να εξετάζει η Επιτροπή κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Δεν έχουν και πόρους άλλωστε για να το κάνουν. Νομίζω ότι είχαμε καταλήξει σε ένα σύστημα δειγματοληψίας για το ποιες θα είναι οι περιπτώσεις που θα εξετάζονται από το σύστημα και ποιες θα χορηγούνται στην Επιτροπή. Προσφάτως δε Μα ζήτησαν να τους χορηγήσουμε πιο πολλέ υποθέσει από μια συγκεκριμένη κατηγορία, όχι το σύνηθε στίγμα. για να επαληθεύσουν την, ε, τον σεβασμό της ανεξαρτησίας μας. Είναι σαφές αυτό, θεωρώ. Προφανώς μπορούμε να εξετάσουμε εκ νέου, αν το επιθυμείτε, τη μέθοδο δειγματοληψίας αν το επιθυμούν, μπορούν να επιλέγουν και αυτοί τις υποθέσεις σε ό,τι αφορά τώρα τον χρόνο εργασίας. Καταλαβαίνω ότι θα μπορούσαν να ερμηνευτούν τα πράγματα όπως μας λέτε, αλλά θα ήταν σίγουρα χρήσιμο να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την διαβίβαση των δεδομένων που ξέρουμε ότι πρέπει να σας χορηγούμε η νομοθεσία είναι πολύ... Δεν διευκρινίζει ακριβώς τι και πώς. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαδικασίες. Ξέρουμε ότι στην τάδε ημερομηνία πρέπει να α, χορηγήσουμε τον κατάλογο των ε, ετησίων εκθέσεων, για παράδειγμα. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να σας πω ότι τρεις νομικές υπηρεσίες ε, στην κοινή του γνωμοδότηση θεώρησαν ότι αυτό θα ήταν απαραίτητο. Δεν είμαι ακόμα πεπισμένος ότι αυτό θα ήταν ε, σκόπιμο να το υπογράψω εγώ ως, ε, ως Ναι. ε, γενικός ευθυντής. Ε, θεωρώ ότι καλά θα κάναμε να συμφωνήσουμε επί του σχεδίου και ελπίζω ο, η, η διαδοχός μου να το υπογράψει σχετικά γρήγορα. ουσιαστικά θα πρέπει να βρούμε κάποιες ρυθμίσεις ρεαλιστικές, ε, κοινή λογική για τις ε, δικαστικέ συστάσεις και το follow-up. Πέρα από κάποιο σημείο το follow-up ε, σε δικαστικές, στις δικαστικές υποθέσεις, το να παίρνουμε τηλέφωνα και να ρωτάμε εισαγγελείς τι έχει γίνει με κάποια υπόθεση δεν αποφέρει πλέον ε, καρπούς γιατί δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση σε ορισμένε περιπτώσεις και δεν έχει και σημασία γιατί τα στατιστικά στοιχεία αυτά δεν θα είναι ποτέ τέλεια. Το βασικό είναι να έχουμε μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει. Περιστασιακά, προφανώς, ε, Πρόεδρε, έχουμε και μια, ε, ένα πραξικόπημα. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν πολλά στοιχεία σε σχέση με τη Ρουμανία, όπου ένας ε, πολιτικός ε, του επαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις ρουμανικές αρχές και οι αρχικές πληροφορίες ε, ξεκίνησαν από δική μας ανάλυση. Άρα προέκυψαν πληροφορίες, ξεκίνησε έρευνα η έρευνα αυτή χορηγήθηκε στις δικαστικές αρχές ε, της ε, Ρουμανίας και η ρουμανική κυβέρνηση ήδη υποσχέθηκε να επιστρέψει 21 εκατομμύρια ευρώ. Και σε μία μέρα η ιστοσελίδα μας δέχεται και πιο πολλές ε, επισκέψεις από ό,τι συνήθως δέχεται σε ένα μήνα, γιατί δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Και συνέβη όμως ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή, γιατί καταδεικνύει το πώς από πλευράς δαπανών και εσόδων μπορούμε να πετύχουμε και μεγάλα αποτελέσματα. Βέβαια, απαγγελία καταγγελιών έγινε, δεν έγινε ακόμα. Ε, δεν έλευθησε η δικαστική απόφαση. Θα πρέπει να γίνει ακριβής ανάλυση για το τι συμβαίνει και σε πιο μικρές ε, υποθέσεις. Ο, η πρόεδρος, ο πρόεδρος επίσης ανέφερε τη σημασία του να εξετάσουμε πότε κλείνει μια υπόθεση, κατά πόσο γίνεται αυτό σωστά. Από όσο θυμάμαι, περίπου οι μισές πληροφορίες από τις λαμβάνουμε ε, δεν εξετάζονται περαιτέρω λόγω έλλειψης αρμοδιότητας και συνήθως είναι σαφές εξ αρχής από τα γεγονότα κατά πόσον υπάρχει αρμοδιότητα του Όλαφ ή όχι. Υπάρχει ένα περιθώριο περιπτώσεων και υποθέσεων, περίπου 100 ας πούμε υποθέσεις, τις οποίες ε, τις ε, ανοίγουμε χωρίς ε, ανάγκη να τις εξετάσουμε σε βάθος, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν τα κριτήρια Κάποιες άλλες υποθέσεις χρειάζονται πιο αναλυτική έρευνα για να διαπιστώσουμε κατά πόσο πληρώνται τα τακτητήρια. Και υπάρχουν και κανένα δυο πάντα στις οποίες σπάζουμε το κεφάλι μας. Ε, αναλογιζόμαστε πόσους πόρους θα χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, τον αριθμό των ε, ερευνητών επιστηρετών επικοινωνιών που μιλούν και την αντίστοιχη γλώσσα. Αν το επιθυμεί η Επιτροπή, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για το ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε και πώς και τι θα πρέπει να εξετάζει η Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να σας δώσω χιλιάδες υποθέσεις να εξετάσετε για κάθε χρόνο. Θα σας καθυστερούσε υπερβολικά. Αλλά ε, από αυτόν των στοιχείων μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις σας προς εμάς πολύ χρήσιμες και ωφέλιμες. Δεν ε, μας ήταν όλες ευχάριστες στο παρελθόν. Δεν θέλαμε να τι ακολουθήσουμε απαραίτητα όλε, αλλά είναι θέμα του προσυζήτηση και μπορεί να είναι επικοδομητική η συζήτησή μα. Ε, κλείνοντας, Πρόεδρε. Νομίζω ότι και από τι δύο πλευρέ. υπάρχει απόλυτη προθυμία να βελτιωθεί αυτή η σχέση και για το μικρό χρονικό διάστημα που θα παραμείνω εδώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το πετύχω αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή είδηση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι για δύο αριθμούς. Για το σύστημα ε, διαχείρισης. Ισχύει αυτό με τα 9 εκατομμύρια και ότι θέλετε άλλα 5 εκατομμύρια. Και μετά πόσο κόστησε η μελέτη εξολόγηση ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα 9 εκατομμύρια είναι πάνω κάτω σωστά, τα 5 εκατομμύρια. Είναι η κασία. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω για τα 5 εκατομμύρια. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω υπεύθυνη απάντηση για το πόσο περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν. Για τη μελέτη, ποια μελέτη ακριβώς εννοείται, αξιολόγηση, evaluation standard. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία. Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, λιγότερο από 400.000, αλλά δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν συμφωνείτε, με mail. Ναι, να το στείλετε, αλλά όλα τα έξοδα παρουσίασης και τα λοιπα πρώτη και 2 Μαρτίου ήταν η μεγάλη εκδήλωση. Θέλουμε το συνολικό κόστος και όχι το μερικό. Γιατί όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Με την όλα αυτά έχουμε ξαναδεί αυτά. Κύριε Μόλτερ θέλετε να απαντήσετε ξανά. Όχι. Δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω αυτά που είπε. Α, συγγνώμη, το διακόπτη, Πρόεδρος. η Υποπτική Επιτροπή έχει θέματα ε, στέγης και ε, έδρας και τα λοιπά. Τι γίνεται. Ε, σας απάντησα σε αυτό. Να τελειώσω όσο πρώτο που σας έλεγα. Έχουμε καλές θέσεις, καλές σχέσεις συνεργασίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε το λεγόμενο working arrangement της διευθετήσεις εργασίας για μια καλύτερη ροή πληροφοριών. Αυτό που ρωτήσατε τώρα για τη μετακόμιση της γραμματείας δεν έχουμε ικανοποιηθεί όλοι, δεν έχουμε δει τα πλέον εκτήματα. Αλλάξαμε κτίριο, καλά είμαστε σε, άλλη δομή, σε άλλο μέρος του κτιρίου. Έχουμε αποκοπή ε, από τις πληροφορίες και δεν έχουμε ακόμα εγκατασταθεί, είναι λίγο πρωτόγονες εκεί ε, οι συνθήκες στέγασης. Δεν έχουμε αίθουσα συνεδριάσεων. Πάνω από έξι μήνες μετά τη μετακόμιση των υπηρεσιών μας, τη δουλειά πάντως την κάνουμε. Στην νομοθεσία εκτός της Όλαφ. Τώρα ολοκληρώνουμε το σύστημα που θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Έχουμε ένα ειδικό καλώδιο από την Όλαφ προς το νέο μας κτίριο, τα νέα γραφεία. Ε, θα έχουμε και επιπλέον ε, υπολογιστές για να έχουμε πρόσβαση ξανά όπως και πριν στο δίκτυο Όλαφ. Αλλά έξι μήνες και πλέον το στερηθήκαμε αυτό και δεν είχαν τρελαθεί όλοι από ενθουσιασμό όταν μετακομίσαμε. Άρα τι να κάνουμε, αλλάξαμε γραφεία και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με επιτυχία. Πάντως το μεγαλύτερο παράπονο είναι ότι η γραμματεία στο κτίριο PMO σημαίνει ότι είναι ξένο σώμα. Εκεί διαχειρίζονται μισθούς, ε, έξοδα νοσηλείας, συντάξεις κλπ. Και όταν είσαι μια μονάδα που θέλεις να συζητήσεις με αμοιδεάτες σου για την πρόοδο, ε, ήταν καλύτερα όταν στεργαζόμασταν στην Όλαφ. Τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σκεφτήκαμε και άλλα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά προς το παρόν γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να τα αλλάξουμε πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Είναι διαδικασία βαριά αυτή, απαιτητική, κάποια στιγμή του χρόνου. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και ε, από το νέο Γενικό Διευθυντή. Αυτή τη στιγμή ε, τα καταφέρουμε εκ των ενόντων, αλλά δεν είναι και τεράστια επιτυχία. Ναι. Και αυτό είναι μία από τις αδυναμίες του κανονισμού, Όλαφ. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμόζουμε την νομοθεσία σε πρόσωπα. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου η νομοθεσία για την εισαγγελία είναι πολύ καλύτερη. Και θα πρέπει να το πω και αυτό στους συναδέλφους. Εμείς που είμαστε αρμόδιοι για τον προπολογισμό, αν δεν καταφέρουμε να στήσουμε με τέτοιο τρόπο ε, μια υπηρεσία που να μπορεί να λειτουργεί καλά και να συνεργαζόμαστε, τότε αυτοί που ασχολούνται με την, ε, τα θέματα της δικαιοσύνης και τα εσωτερικά θα μας στριμώξουν πάρα πολύ. Αν δείτε τι γράφει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πραγματικά θα εκπλαγείτε, γιατί όταν ασχολούνται αυτά, με αυτά τα θέματα εκείνη που είναι της δικαιοσύνης και των εσωτερικών ε, και λιγότερο εκείνη των οικονομικών, βλέπουμε τι συμβαίνει. Πάντως, ε, με αυτά που άκουσα σήμερα τα βρίσκω πολύ ενθαρρυντικά και στη δεύτερη γνωμοδότηση, αυτά που λέει η Εποπτική Επιτροπή, έχει προτάσεις για το μέλλον, για μεταξέλιξη κτλ. Χρειάζεται δουλειά εδώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να σα ευχαριστήσω και εσάς και την Επιτροπή και την Εποπτική, όλο το επιτελείο σας. Θα παραμένουμε σε επαφή όπως πάντα. Ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 15 στην ημερήσια διάταξη. Έκτακτη ε, έκθεση για ε, ελέγχου στην Αλία. Από το ελεκτικό συνέδριο θα μας μιλήσει ο κύριος Βόιτσεκόφσκι, ε, δικός μας ε, εισηγητής είναι ο κύριος Τσέλε. Κύριε η φεστιβάλ σήμερα δικό σας είναι η συνεδρίαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω την επόμενη εκθεσή μας με τίτλο Ευρωπαϊκή έλεγχοι στην αλληλεία χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Όπως ξέρετε, στόχος της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής είναι να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και της αλληλείας αλλά και των αποθεμάτων. Υπάρχει υπεραλίευση, άρα χρειάζονται και άλλες προσπάθειες έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε με ε, αποτελεσματικό τρόπο και βιώσιμο ε, τα αλληλεύματα. Τι μας ζητήθηκε να ελέγξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σύστημα ελέγχου αποτελεσματικό για την αλεία. Η απάντηση είναι όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούμε να σας πούμε ότι είμαστε στη μέση μιας προσπάθειας, στη μέση του δρόμου. Ε, σωστή κατεύθυνση μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο τέρμα διότι από την περασμένη μας ε, ε, εργασία το 2007 που είχαμε κάνει τον έλεγχο, έχει βελτιωθεί σημαντικά το σύστημα ελέγχου την τελευταία δεκαετία, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια, αλλά τα μέλη που δεν είχαν ακόμα εφαρμόσει πλήρως ε, τους κανονισμούς για τον έλεγχο και κάποιες διατάξεις χρειάζονται να κάνουν αλλαγές. Ποια ήταν τα κύρια ευρήματα. Πρώτον, μια στιγμή να τα βρω τα ευρήματα. Πληροφορίες για το στόλο. Για αποτελεσματικό έλεγχο θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο αλευτικός στόλος. Με αξιόπιστες ε, πληροφορίες και στοιχεία. Στα κράτη-μέλη που επισκεφτήκαμε, τέσσερα τον αριθμό, τα οποία είναι σημαντικά τα μεγαλύτερα έτσι, αλλιευτικά κράτη που έχουν το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο. Ε, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι οι τέσσερις χώρες που επισκεφτήκαμε. Αυτοί δεν ε, ελέγχουν αποτελεσματικά τη χωρητικότητα του στόλου, ε, τα νεολόγια κτλ τα τέσσερα κράτη-μέλη δεν ελέγχουν τη χωρητικότητα σε τόνους των αλληλευτικών του σκαφών, ενώ δύο από τα τέσσερα κράτη δεν είχαν ακόμα προχωρήσει ε, στις απαραίτητες ε, ε, διευκρινήσεις και επαληθεύσεις το, της ισχύω του κινητήρα των σκαφών. Και υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στα όσα γράφουν τα νεολόγια ως καταχώρηση και ε, όσα γράφουν τα συνοδευτικά έγγραφα ε, των σκαφών των ίδιων. Αυτά είναι για το στόλο. Άλλο έβριμα. Τα μέτρα διαχείρισης. Ε, διαπιστώσαμε ότι γενικά τα κράτη-μέλη ελέγχουν όταν αντιρούνται μάλλον τα μέτρα αυτά. Έχουν ένα σύστημα VMS, ε, μια τεχνολογία δορυφορική για τον εντοπισμό και την ανείχνευση ε, των σκαφών και την παρακολούθησή τους. Λειτουργεί καλά αυτό το σύστημα, αλλά 89% του ελευτικού στόλου δεν εντάσσεται στο VMS. Δεν παρακολουθείται από το σύστημα το δορυφορικό. Αυτό βέβαια αφορά τα μικρότερα σκάφη τα υπόλοιπα που παρακολουθούνται, το 11% είναι τα μεγαλύτερα σκάφη που αλλιεύουν τα περισσότερα, τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό. 89% των μικρών αλλιευτικών σκαφών δεν παρακολουθούνται με το δορυφορικό σύστημα. Μετά, ε, επόμενο έβριμα. Έχουμε το πρόβλημα ε, του, της απονομής ε, ποσόστοσης. Τα κράτη-μέλη που επισκεφτήκαμε ε, απορροφούν ε, την ποσόστοση που τους έχει ανατεθεί. Όταν όμως αναθέτουν σε οργανώσεις αλλιέων να κατανείμουν τις ποσοστώσεις, δεν ξέρουμε ποια κριτήρια το κάνουν αυτές οι οργανώσεις αλλιέων και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Αυτό σημαίνει αδιαφάνεια και αυξάνει τον κίνδυνο να εξυπηρετούνται ειδικά συμφέροντα ορισμένων οικονομικών παραγόντων εις βάρος κάποιων άλλων. Επόμενο εύρημά μας. είναι τα στοιχεία και τα δεδομένα για τις αλληλευτικές δραστηριότητες που συλλέγονται ε, στα πλαίσια του κανονισμού ελέγχου δεν είναι αρκετά αξιόπιστα ούτε αρκετά πλήρη. Η διαδικασία ε, επικύρωσης των δεδομένων αυτών των στατιστικών στοιχείων στα κράτη-μέλη είναι ανεπαρκής, μη ικανοποιητικές και υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα ε, στις συνολικές ποσότητες ε, της αλήφθησης που διαθέτουν ως στοιχεία τα κράτη-μέλη και όσα διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία από τη στιγμή ε, ε, των δηλωμένων εκφορτώσεων ε, και της πρώτης πώληση. Μετά, το σύστημα επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων ελέγξαμε επίσης. Και τι διαπιστώσαμε. Θα πρέπει η κύρωση να συνδέεται ε, με την παράβαση και το οικονομικό συμφέρον. Στην Ισπανία αυτό γίνεται συστηματικά, στη Σκωτία λιγότερο. σε κάποιες περιπτώσεις ε, προβλέπεται αυτό από την νομοθεσία στην Ιταλία και στην ε, Γαλλία, αλλά δεν εφαρμόζεται πάντα στην πράξη. Στη σελίδα 48 της έκθεσής μας έχουμε πληροφορίες για την δραστηριότητα των επιθεωρήσεων. Δείχνει ότι γίνεται στην Ισπανία τρία χρόνια διήρκησε ο έλεγχο. 2014, μάλλον 13 διορθώνει ο μιλητή, από το 2013 μέχρι το 2015, στην Ισπανία πάνω από 23.000 έλεγχοι έγιναν επιθεωρήσεις, στη Γαλλία περίπου 40.000, στην Ιταλία 18.000, στο Ηνωμένο Βασίλειο 16.000. Ε, διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις στην Ισπανία, ας πούμε, 4.700, στην Ιταλία 3.500. Δείχνει αυτό ότι είναι σοβαρές οι επιθεωρήσεις που γίνονται και εμπεριστατωμένες, εν πάση περιπτώσει, και στοχευμένες για να ε, εντοπίζουν τις παρατυπίες και τα προβλήματα. Αλλά το θέμα είναι, είναι αρκετά αποτρεπτικές οι που επιβάλλονται. Γιατί είδαμε πολλές περιπτώσεις και σκαφών όπου τιμωρούνται πέντε φορές σε μία τριετία και συνεχίζουν να παρανομούν. Άρα το σύστημα επιβολής κυρώσεων ούτε αποτρεπτικό είναι ούτε αποδίδει. Αυτά ήταν τα βασικά ευρήματά μας και οι συστάσεις μας τώρα οι βασικές είναι αυτές που βλέπετε. Να επιβάλλουμε αποτρεπτικές ε, κυρώσεις ιδιαίτερα για παραβάσεις κατ' εξακολούθηση να εφαρμόζεται πλήρω το point system. Πολύ σημαντικό αυτό. Με επινές ε, να αφαιρούνται πόντι, δεν εφαρμόζεται πλήρω στην πράξη. Ένα σύστημα ανταλλαγής προφοριών για τις ε, παραβάσεις και τις κυρώσεις. Βελτίωση των στοιχείων, βελτίωση εξακρίβωση των στοιχείων, ιδιαίτερα για τα μικρά σκάφη promote electronic Ηλεκτρονικές δηλώσεις για μικρά σκάφη. Μέτρα διαχείρισης επίσης να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύστημα κατανομής των ποσοστώσεων για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Ένα σύστημα εναλλακτική εντοπισμού των μικροτέρων σκαφών, εξακρίβωση των στοιχείων στον ιολόγιο και προτείνουμε και κανόνες για την εξασφάλιση και την εξακρίβωση της χωρητικότητας. Ε, αυτά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσέλε, ο οποίος είναι ο εισηγητής της Επιτροπής σας, γιατί στο έγγραφο εργασίας του υποστηρίζει τις δικές μας συστάσεις. Καμιά φορά ε, ε, τις βρίσκει και υποβοηθητικές και ενισχύουν το κείμενο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία κυρία Πρόεδρε να σας παρουσιάσω την παρούσα έκθεση που είναι σημαντική πιστεύω για να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το σύστημα ελέγχου στην αλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφος Τσέλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βοητσεχόφσκι και τους συνεργάτες του από το ελεγκτικό συνέδριο. Πώς ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, αφού υπάρχει ειδική έκθεση για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ε, εταιρικών ε, συμβάσεων για την αλληλεία, ασχολήθηκαν και με το συγκεκριμένο θέμα για το εσωτερικό πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι αυτά που λέγει και διαπιστώνει το ελεκτικό συνέδριο ανταποκρίνονται στις δικές μας ανησυχίες και φόβους και δεν διασκεδάζονται καθόλου αυτές οι ανησυχίες. Απομένει πολλή δουλειά. Το ψάρι είναι από τα πιο αγαπημένα τρόφιμα και συνιστάται ως υγιεινό τρόφιμο. Αυξάνονται ε, τα αλλιεύματα, η αλήψη δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα διαβάζουμε διάφορες εκθέσεις και επιστημονικά στοιχεία βλέπουμε που λένε ότι μειώνονται τα αλλιευτικά αποθέματα. Γι' αυτό καλό ήταν που επικεντρώθηκε το ελεκτικό συνέδριο σε κράτη-μέλη που από μόνα τους ε, έχουν το 50% του αλλιευτικού στόλου και ε, αλλιεύουν στο Βόρειο Ατλαντικό αλλά και στη Μεσόγειο. Φέτος τον Απρίλιο βγήκε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλεγε ότι 93% όλων των ε, αλλιευμάτων, όλων των ειδών στη Μεσόγειο απειλούνται ε, με οξύ τρόπο και αν δεν λάβουμε μέτρα στην, ε, την επόμενη γενιά η Μεσόγειος θα έχει μόνο αχινούς, πλαστικά απόβλητα και ε, έδουσε αυτά από περιεκτικότητα στη Μεσόγειο. Ε, άρα χρειάζεται έλεγχο. Το, το σύστημα VMS, όπως είπε και ο κύριος Βοτζεκαυσκή, καλύπτει μόλις το 11% του ελευτικού στόλου, αλλά 89% ανεξέλεγκτα ε, μπορούν να ψαρεύουν. χωρίς βιώσιμο έλεγχο για το τι αλλιεύουν και με ποιο τρόπο. Επίσης, ε, είπε ο κ. Βοητσοχόφσκι ότι η ποιότητα των δεδομένων είναι διαφορετική. Τα συστήματα που συλλέγονται ε, σημειώνεται η χωρητικότητα και ισχύς ε, μάλλον η ισχύ των ε, κινητήρων, αλλά όχι η χωρητικότητα, η ερευτική δυνατότητα των σκαφών και η ε, εκφόρτωση των ποσοτήτων στα διάφορα κράτη-μέλη. Στα διάφορα κράτη-μέλη επίσης έχουν τις ποσοστώσεις τις οποίες διαχειρίζονται κάποιοι οργανισμοί και τις αναθέτουν σε αλληλείς ε, με αδιαφάνεια τελικά. Ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, ποιος μοιράζει τις ποσοστώσεις και ποιος τις κατανέμει. Και είναι αυτή η δίκαιη κατανομή σε όλους τους ε, ψαράδες και τέτοια πράγματα. Κάτι άλλο δεν θα πω ότι είναι γελίο, είναι περίεργο. Την περασμένη εβδομάδα κάνανε ερώτηση οι συνάδελφοι της Επιτροπής Αλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι προτίθεται να πράξει έτσι ώστε οι Ποσειδονίες στη Μεσόγειο να μην μειώνονται. Λες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπάλληλοι εκεί της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ να, φυτεύουν υποβρύχια λιβάδια. Εδώ έχουμε ρημάξει ε, τη θάλασσα, χτίζουμε μαρίνες και ε, οργιάζει η ε, ερασιτεχνική αλία από σκάφη αναψυχής και διάφορα άλλα ιστιοπλαϊκά κλπ. Οπότε δεν χρειάζεται να εκπλησώμεθα όπου μειώνονται τα αλλιεύματα και με τρόπο μάλιστα εντυπωσιακό. Οι Ποσειδονίες, ξέρουμε, ότι έχουν και πολύ μεγάλη σημασία για τα ε, ψάρια, για να μεγαλώνουν από ε, γόνοι, να γίνονται ενήλικα. Κάνει προτάσεις στο ελεκτικό συνέδριο για τη βελτίωση του συστήματος. Ε, πήρα το θάρρος από πλευράς μας να κάνω και εγώ κάποιες προτάσεις. Το σύστημα παρατήρησης των σκαφών θα πρέπει να επεκταθεί όχι μόνο στα μεγάλα σκάφη, αλλά και σε καΐκια μεγέθους 12 με 15 μέτρα. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο σύστημα VMS. Ξέρω ότι εδώ υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αλλά και για λιγότερο από 12 μέτρα κάποια συστήματα εντοπισμού και ανείχνευσης θα πρέπει να υπάρχουν μικρότερα και φτηνότερα. Όπως λέει και μια ρωσική παροιμία όμως, ε, καλή εμπιστοσύνη, αλλά καλός και ο έλεγχος. Ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη, αλλά ακόμα πιο αναγκαίος είναι ο έλεγχος. Συλλογή στοιχείων. Δεν είναι ηλεκτρονική, είναι στα χαρτιά. Αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί και να ε, μεταβληθεί το σύστημα σε ηλεκτρονικό για σκάφη και κάτω των 10 μέτρων, έτσι ώστε τα συστήματα να είναι συμβατά για να ανταλλάσσουν πληροφορίες στα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υποπτίας της πράγμα που είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα πόρισματα του ελεκτικού συνεδρίου και θα πρέπει σταδιακά να ε, εισαχθούν νέα συστήματα υποχρεωτικής ε, αξιόπιστης αναφοράς και για μικρά σκάφη κάτω των 10 μέτρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό και τα όσα αυτός ορίζει. Και πραγματικά έχει έρθει η ώρα να ελεγχθεί ο κανονισμός για τα αλλιεύματα, να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα μέτρα και όπου χρειάζεται να επεκταθούν. Αλλά κυρίως να φροντίσουμε και να προσέξουμε τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόζουν όλα αυτά και μάλιστα με τον τρόπο που ορίζουν τα κείμενα του κανονισμού. Κατά τα άλλα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα είναι μια τρύπα στο νερό. Και κάτι άλλο που έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε στη στρατηγική για το 2020 είναι να φροντίσουμε φορεία και βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας. Και αν μη τι άλλο, σε ό,τι αφορά την αλία, αυτό δεν τηρείται πάντα. Άρα στρεφόμαστε και κατά τον ιδρύμα μας τον στόχο και τους παραβιάζουμε. Ευχαριστώ και πάλι το ελεγκτικό συνέδριο που επιλήφθηκε του θέματος αυτού και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια και έχουμε και κάποια πιο συνεπή στάση απέναντι στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή κάποιων νομοθετημάτων τα οποία από κοινού αποφάσισαν και δεσμεύτηκαν να είναι πιο συνεπείς στην εφαρμογή και να ληφθεί υπόψη φυσικά στην διαδικασία αυτή και η δική μας σύσταση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ήθιστε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, πριν πάρει το λόγο ε, ο, η Κομισιόν, <laughs> δίνουμε πάντα το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ. Α, φαίνεται ότι δεν μου τα είπε καλά η Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, να, θα πάρετε το λόγο και θα δώσω... Ε, στην, θα μείνει για την Κομισιόν λιγότερος χρόνος, αλλά θα τα καταφέρει ο κύριος Αλαφράγκα και μετά. Ε, η κυρία Γιάννα Σέντερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Ε, θα διαβάσω τις ε, σημειώσεις του κυρίου Μανσούρ που είναι ο σκιώδης μας και δυστυχώς μετά πρέπει να φύγω. Εν πάση περιπτώσει θα μου πούν οι βοηθοί της ομάδας τα σχετικά. Ε, ζητά συγγνώμη ο σκιώδης μας που δεν μπορεί να είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστεί τον κύριο Ζέλερ για την εργασία του, ε, καθώς επίσης ε, και τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την παρουσίαση του. Ε, συμφωνούμε ότι πραγματικά από το 2000, για, για, το, το 2019 θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των κανονισμών ελέγχου της αλίας, γιατί πολλές παράμετροι έχουν πλέον αλλάξει. Υπάρχει και μία παράμετρος που δεν είναι έχει ληφθεί υπόψη ε, είναι αυτή της κλιματικής αλλαγής που όμως ε, έχει πάρει πολύ σοβαρές ε, διαστάσεις και δημιουργεί πρόβλημα και στην θαλάσσια πραγματικότητα γενικότερα αλλά και στην παράκτη ειδικότερα. Η ελεία είναι σημαντικό στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά βεβαίως όπως είπε και ο κύριος Ζέλερ αποτελεί πολύ υγιεινή διατροφή η ισορροπία ανάμεσα στην αλλιευτική δραστηριότητα και τους αλλιευτικούς πόρους και την διατήρηση των οικοσυστημάτων και της ε, χλωρίδα, της πανίδας είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ε, επίσης, το γενικό πλαίσιο ελέγχου της αλίας πέρα από το ότι ε, ο κανονισμός είναι κανονισμός ε, ελέγχου, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις ε, λόγω διαφοροποιημένης εφαρμογής των αρχών και λόγω των διαφορετικών εστιάσεων που κάνει η κάθε χώρα και που έχουν εθνικό χαρακτήρα η ανταλλαγή στοιχείων και βελτίστων πρακτικών, όπως ε, άλλωστε το αναφέρει και το Ελληνικό Συνέδριο, ε, πρέπει να ε, διευρυνθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων πραγματικά αξιόπιστες αλλά και ταυτόχρονα διαφανείς. Η τεχνικές ε, εντοπισμού δίνουν βεβαίως ε, ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία, διευκολύνουν ε, τον έλεγχο των σκαφών πάνω από 15 μέτρα, αλλά για τα μικρότερα σκάφη, μικρότερα από 12 μέτρα, δημιουργούν προβλήματα Ε, είτε γιατί ο εξοπλισμός ε, είναι πολύ ακριβός, ε, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ μικρών σκαφών βιοτεχνικής αλληλείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναλογικότητα. Όσον αφορά τις κυρώσεις, ε, το γεγονός ότι αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, οδηγεί ε, σε μεγάλες διαφοροποιήσεις, αν όχι στρεβλώσεις. και ε, άλλωστε και στην έκθεση του ελεκτικού δικαστηρίου προκύπτουν συνεδρίου ε, προκύπτουν ε, ε, διαφοροποιήσεις, έλλειψη αναλογικότητας και εν πάση περιπτώσει εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο καλύτερο για τις κυρώσεις και μάλιστα θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα και να υπάρξει μια εναρμόνιση των κυρώσεων έτσι ώστε να υπάρχει ή αντιμετώπιση. Ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάποιο στοιχείο ε, το οποίο μας ε, προβληματίζει όλο και περισσότερο. Είναι το θέμα της παράνομης αλίας από εθνική σκάφη, από ευρωπαϊκά σκάφη, αλλά όλο και περισσότερο και μάλιστα με βιομηχανικό τρόπο ε, ε, γίνεται από ε, σκάφη τρίτων χωρών, ακόμα και από χώρες οι οποίες έχουν διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, ας πούμε, μια περίπτωση, την περίπτωση της Παπρετανίας που την αναγνωρίζουν όλοι και τη γνωρίζουν όλοι. Όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της αρμοδιότητας αυτών των τρίτων χωρών ε, όπως η Κίνα ας πούμε ή όπως ε, η Ιαπωνία οι, οποία, ε, οι οποίες δεν σέβονται κανένα κανόνα και οι οποίες δεν υφίστανται κανέναν έλεγχο. Ε, ε, ελπίζουμε ε, και ευχόμαστε κάποια στιγμή σε κάποια έκθεση του το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει μια αναφορά. Γιατί αν δούμε το, την γενικότερη εικόνα όλου του τομέα ε, νομίζω ότι μπορούμε ε, να, ε, να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε υπερβολικούς κανόνες για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα ανοίγουμε το δρόμο για αθέμητο ανταγωνισμό με, σε σκάφη τα οποία τα οποία ε, αλλιεύουν χωρίς να σέβονται κανόνες ε, με τρόπο άναρχο και ε, παράνομο. Θα θέλαμε λοιπόν, επειδή υπάρχει, προκύπτει μεγάλη στρέβλωση του ανταγωνισμού με τον τρόπο αυτό, θα θέλαμε λέω να μας δώσει κάποια στιγμή το ελεγκτικό συνέδριο τη συνολική εικόνα και όχι μονάχα ε, μια εικόνα σχετικά με τις ακυρώσεις ή την εικόνα των ελέγχων για την ευρωπαϊκή Αλία αποκλειστικά και μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαλαμάνκα, θα είμαι πολύ σύντομος κυρία Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω ε, με την κυρία Αγιάλα ε, και θα πω και εγώ ότι η εργασία του κυρίου Ζέλερ είναι πάρα πολύ καλή. Διάβασα το προσχέδιο του εγγράφου εργασίας και δεν ξέρω αν κάπου έχει προκύψει κάποιο λάθος ή αν είναι πραγματικά ε, η θέση του εισηγητού. Στο σημείο 1 αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υποβάλλει ε, κάποιες προτάσεις 2019-2020 και στο τέλος λέει ότι για να βελτιωθεί η ελευτική ικανότητα τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι το 2018 δεν ξέρω, όσο κι αν ε, είμαστε γρήγοροι και, τα, και ταχύτατα εγκρίνουμε την εργασία του, είμαστε ήδη 21η Νοεμβρίου του 2017. Δεν ξέρω εάν ε, ξέφυγε το λαθάκι αυτό ή εάν πραγματικά θέλει ε, να πιέσει χρονικά την κατάσταση. Και όσον αφορά την Κομισιόν, πριν δώσετε το λόγο κύριε Πρόεδρε στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, θα ήθελα να μάθω το εξής. Ποια είναι τα χρονικά περιθώρια τα οποία ε, προβλέπετε για τον ε, ελεγκτικό κανονισμό. Μα ε, μας λέει το έγγραφο ότι η Κομισιόν δέχεται εν μέρη ε, κάποιες προτάσεις αλλά δεν έχει πάρει απόφαση αναθεώρησης του κανονισμού. Αλλά βεβαίως πριν αναθεωρηθεί ο κανονισμός θα πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση κλπ. Και βεβαίως ε, ε, ε, έλεγχος τη επίπτωση των προτινομένων μέτρων. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μας δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα λοιπόν να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, πάντα το ερώτημα είναι φυσικά ποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή. Μάλιστα, βλέπω ότι κάποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πολύ ωραία. Ε, Καλό απόγευμα. Ε, λέγομαι Φρανσίσκα Ρένα και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, ε, το Ελληνικό συνέδριο, να το ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, γιατί επανειλημμένα είχαμε την ευκαιρία ε, να ευχαριστήσουμε το ελληνικό συνέδριο για την έκθεσή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την πολύ πιστή έκθεση του εισηγητού κυρίου Ζέλερ πιστή λέω όσον αφορά τα συμπεράσματα του, της εκθέσεως ε, της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μας παρέχει μια σωστή ε, ανάλυση της κατάστασης την στιγμή ακριβώς του οικονομικού ελέγχου, του audit. Ε, τότε δηλαδή, τη στιγμή που έλαβαν χώρα στις ε, χώρες μέλη αυτή η έλεγχη και βεβαίως μπορούμε απολύτως να συμφωνήσουμε με τα συμπεράσματα. Δηλαδή, ε, παρά το γεγονός ότι πολλά έγιναν τα τελευταία χρόνια, χρειαζόμαστε ακόμα περαιτέρω πρόοδο γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ κρίσιμα ερωτήματα όσον αφορά τον έλεγχο κυρίω, που αποτελεί ούτως ή άλλως τη σπονδυλική στήλη των πολιτικών της ε, ε, Ένωσης. Ε, πρέπει να πω ότι έχουμε διαρκείς εξελίξεις, διαρκείς βελτιώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και χάρη στην δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ήδη έχουμε ταυτοποιήσει μια σειρά ε, δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα ε, και στις χώρες που έχουν ελεγχθεί και σε άλλες χώρες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις οι οποίες έχουν αναφερθεί. Επομένως η διαδικασία είναι διαρκής, οπωσδήποτε θα συνεχίσει όπως άλλωστε ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Επίσης και παρομοίως η παρούσα, ε, ο παρόν κανονισμός ελέγχου δεν είναι ο πλέον προσήκον ε, και αυτό σε πολλά πεδία δεν δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις σε όλα τα τμήματα ε, των, των στόλων. Παράδειγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό των μικρών σκαφών. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις όσον αφορά τις διατάξεις αυτού του κανονισμού ελέγχου. Θα ήθελα ε, επίσης να συμφωνήσω με αυτό ε, που αναφέρθηκε από τον τελευταίο παρεμβαίνοντα, δηλαδή ε, να ξεκαθαριστεί το, το περιεχόμενο του κανονισμού ελέγχου, γιατί η Κομισιόν είχε δεχτεί όχι πλήρως και με κάποιες επιφυλάξεις τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο λόγος είναι απλός. Τη στιγμή που ψηφίστηκε, που, που συζητήθηκε η έκθεση αυτή, η Κομισιόν δεν ήταν ακόμα σε θέση τα Μεταβεβαιότητος να δώσει ε, σαφείς ενδείξεις όσον αφορά την προσαρμογή ε, της ε, οδηγίας, συγγνώμη, του κανονισμού. Η διαδικασία όμως πλέον έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία μελέτης επιπτώσεων του νέου κανονισμού και βάσει των παρόντων σχεδιασμών ε, εντός του Απριλίου 2018 θα έχουμε ε, το ε, σχέδιο του κανονισμού. Είναι προφανές ότι όλες οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα ληφθούν υπόψη και μάλιστα με τρόπο απολύτως λεπτομερή στην σύνταξη και εκπόνηση του νέου κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι ε, κατά την άποψή μας ε, είναι απολύτως χρήσιμες οι συστάσεις και γενικότερα η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι λέω απολύτως χρήσιμες ε, στην Κομισιόν. Ε, αναφέρομαι ε, ε, επίσης και στα συμπεράσματα, της προτάσεις οι οποίες αφορούν την επιτήρηση, οι οποίες αφορούν την αξιοπιστία των στοιχείων που αφορούν τα αλλιεύματα και όσον αφορά τα τονάζ λοιπά και την ισχύ των κινητήρων. Βεβαίως, μην περιμένετε ότι θα υπάρξει επανάσταση στο σύστημα ελέγχου. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η υλοποίηση των μέτρων είναι εξαιρετικά ε, σημαντική ότι ένα μεγάλο μέρος των πόρων που χρησιμοποιεί η Κομισιόν αφιερώνονται ε, ακριβώς στην ε, υλοποίηση ε, των μέτρων από πλευρά των κρατών μελών και ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και βάσει ακριβώς και χάρη στα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέγει Πρόεδρος. Κύριε Ζεχόφσκι, θέλετε και, και, θέλετε και εσείς να πάρετε το λόγο. Εν συντομία να χρησιμοποιήσω και την πολωνική γλώσσα. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και την ε, Επιτροπή Ελέγχου του και θέλω να πω ότι ήταν πολύ καλή η συνεργασία με την Επιτροπή και καλή ήταν η κατανόηση επίσης ότι αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της επιθεώρησης. Αυτό καταδεικνύει ότι παίρνουν τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά και τις συστάσει μας, σε ό,τι αφορά και την σύσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Αλία. Επίσης, όταν παρουσιάσαμε τα πορίσματα και σε ένα ανακοίνωση τύπου, συναντηθήκαμε και με εξωτερικούς φορείς, με εκπροσώπους των ενώσεων και οργανώσεων αλίας, με περιβαλλοντικού και σε οργανώσεις και όλοι εξέφρασαν την επιθυμία να ενισχυθεί το σύστημα. Όλοι καλωσόρισαν τις συστάσεις μας, ενδεχομένως να μην ήταν όλοι ικανοποιημένοι με τα πορίσματα. Όλοι θα θέλαμε καλύτερα πορίσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι συστάσεις έγιναν ευρέως αποδεκτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την κυρία Γελασέντερ και τον κύριο Σαλαφράγκα για τα λόγια αποδοχής των πορεσμάτων αποτελεί πρόβλημα ομολογμένως ότι οι αλλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την χάνουν ίσης αντιμετώπισης και το σύστημα επιβολής κυρώσεων στα κρατημέλη είναι διαφορετικό. Θα ήθελαν προφανώς να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, άρα οι ίδιοι κανόνες είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και Υπάρχει και το θέμα των αλλιευμάτων το οποίο ανέφερε η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Το θέμα των τρίτων χωρών δεν το εξετάσαμε γιατί εξετάσαμε το σύστημα παρακολούθησης των κρατών μελών. Αυτό όμω αποτελεί ένα σχόλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως να χρειάζεται ανάλυση το πρόβλημα αυτό σε ό,τι αφορά τις παράνομες αλλιεύσεις από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και νομίζω ότι στο σημείο αυτό η δουλειά μας θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της κοινής αλληλευτικής πολιτικής και σε καλύτερα αποτελέσματα. Βιώσιμη διαχείριση στη τελική ανάλυση των αποθευμάτων αλληλευμάτων, τα οποία και καλούμαστε να προστατεύσουμε. Κλείνοντα και ο συνάδελφο Τσέλερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα επαναλάβω ότι δεν αρκεί πλέον η εμπιστοσύνη. Εδώ χρειαζόμαστε πλέον ελέγχου. Ιδάλω, ο όλο κανονισμό και η όλη νομοθετική διαδικασία γελιοποιείται. Για μια βιώσιμη λοιπόν ε, αλία χρειάζεται αυτό μετά και από τα απορίσματα του Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και από άλλες εκθέσεις διαπιστώνουμε ότι κάτι θα πρέπει να συμβεί πλέον και γι' αυτό αναφέρω ετήσια στοιχεία για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Σαλανφράγκα. Το έγγραφο εργασία ήταν αρχές Οκτωβρίου έτοιμο και ξέρω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειαζόμαστε χρόνο σε περίπτωση που τα κρατημέλη πρέπει να εφαρμόσουν τον ήδη φυστάμενο κανονισμό το ε, 2018, όπου μιλάμε για προσαρμογή όπου χρειάζεται πιο πολύ χρόνο. Έβαλα 2019 και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είπε ότι ήδη επεξεργάζονται αλλαγή του σχετικού κανονισμού ελέγχου. Και γι' αυτό λοιπόν στο σημείο αυτό διευκρινίσα ως ημερομηνία στόχο το 2020. Σε αυτά τα χρονικά όμως ε, στοιχεία, σε αυτές τις χρονικές στιγμές θα πρέπει να συμβεί κάτι. Και τα αποτύπωσα όλα αυτά λοιπόν στο έγγραφο εργασία. Ιδάλω δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Και ίσω και να κοροϊδεύουμε έτσι και του αλληλεί, οι οποίοι μπορεί τώρα κάτι να βγάζουν από τη θάλασσα ακόμα. Αλλά οι μελλοντικέ γενιέ τι θα έχουν να ψαρέψουν πέρα από ε, πλαστικά σκουπίδια και μέδουσες. Αυτό που ζήτησε η συνάδελφος Αγελά Σέντερ να ελεγχθούν και οι άλλοι που ψαρεύουν στα νερά μας και ενδεχομένω ψαρεύουν και παράνομα. Αυτό το διαπιστώνουμε αν έχουν ένα πιστοποιητικό και αυτοί που ψαρεύουν νόμιμα. Αυτό δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Έχουμε λοιπόν το στόλο, έχουμε το σύστημα παρακολούθησης, αλλά κατά 89% δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό. Και έτσι δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των νόμιμων και παρανόμων αν βελτιώσουμε το δικό μας σύστημα αλλιεύσης ε, και την υποχρέωση πιστοποίησης στο σύστημα επιτήρησης, τότε θα καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά και την παράνομη αλληλεία στα δικά μας τα νερά. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλαφράγκα και πάλι ευχαριστώ Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τσέλερ για τη διευκρίνηση. Είναι πάρα πολύ λογικά αυτά που λέει και ίσως στη γραμμή των όσων μας προτείνει ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση για να βελτιωθεί η βελτίωση, να βελτιωθεί μάλλον η ακρίβεια των τα κράτη-μέλη θα όφυλαν ήδη από τώρα εφαρμόζοντας την κείμενη ε, νομοθεσία να προχωρήσουν ε, σε αλλαγή κτλ. Γιατί όσο και να τρέξουμε δεν προλαβαίνουμε μέχρι το 2018 και όπως εξήγησε ο εισηγητής, πρόκειται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Δηλαδή, για να είμαστε και πιο σωστοί και πιο αυστηροί, να μην βάζουμε στόχους και χρονικούς ορίζοντες που δεν μπορούμε να τηρούμε, αλλά να εφαρμόζουμε και να υλοποιούμε τα ήδη ισχύοντα. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλό θα ήταν να ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά βιώσιμα και αηφόρα. Είναι δύο θέματα που δεν ασχολούμαστε με αυτά ως θα οφείλαμε και με τη συχνότητα ε, που θα έπρεπε. Αλληλεία λοιπόν και γεωργία και ανάψη χρυπέθρου και να κάνουμε καμιά ακρόση και για αυτά τα θέματα και όχι μόνο για διάφορα γενικά και αόριστα και με αυτές τις δαπάνες να ασχοληθούμε. Τελειώνει εδώ η δημόσια συνεδρία. Σε ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να πω ότι έχουμε και μια προκατακτική για το διάλογο όλα την, την ερχόμενη πέμπτη το απόγευμα και κλεισμένο το θυρών και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην προετοιμασία αυτή για την ερχόμενη πέμπτη με χαρά είστε προσκεκλημένοι. Και ποιος δεν έρθει την πέμπτη δεν χρειάζεται τώρα να μείνει. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Λήξη συνεδρίαση.